Uh, uh, Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ, θα προσθέσουμε και λίγο χρόνο για να συμμαζευτούμε. Έχουμε πολλούς να ακούσουμε όμως. Άρα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το βέλτιστο δυνατό τρόπο τον διαθέσιμο χρόνο. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Uh, Καλησπέρα. Είμαι ο Μάλκομ Χάρμπορ. Έχω το προνόμιο να έχω εκλεγεί πρόεδρο τη Επιτροπή Εσωτερική Αγορά και Προστασία Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι μέλο τη βρετανική αντιπροσωπεία, ανήκω στο συντηρητικό κόμμα και έχω ασχοληθεί επί 10 χρόνια με θέματα εσωτερική αγορά. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Επίσης είναι προνόμιο για μένα να μπορώ να καλωσορίσω πολλούς συναδέλφους βούλευτες από κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που ήρθαν για ανταλλαγή απόψεων, για να συνομιλήσουμε με θέμα τη σημαντικότατη αυτή πρόταση για τις καθυστερήσεις πληρωμών και τον ανασχεδιασμό της σχετικής προτάσεως. Ήδη είδαμε κάποιες προτάσεις σας και είναι πραγματική δυνατότητα αυτή που έχουμε να συναντηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο και να μπορέσουμε να σα ακούσουμε. Και βεβαίω, σύμφωνα με τι διατάξει συνθήκη τη Λισαβόνο, η επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια θα ενισχυθεί σημαντικά. Αυτή η Επιτροπή θεωρώ ήταν ε, πάντα στην πρώτη γραμμή αυτών των θεμάτων. Είχαν επιτυχέστατη συνεδρίαση όσον αφορά τα οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην προηγούμενη θητεία και αυτή είναι η πρώτη δυνατότητα που έχουμε έκτοτε μετά τις εκλογές να ξανασυναντηθούμε. Και ίσως θα θέλατε να γνωρίζετε και απευθύνομαι προς τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων λέγοντας αυτό ότι στις 17 και 30 μετά την λήξη της συνεδριάσεώς μας θα διεξαχθεί η πρώτη βίντεο διάσκεψη με την Επιτροπή Δικαιωμάτων Καταναλωτών της Assemblée Nationale της Γαλλικής Εθνοσυνελεύσεως. Όποιος θέλει να δει πώς λειτουργεί είστε ευπρόσδεκτοι ως θεατές. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της προσπαθίας να έχουμε στενότερη επαφή με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κάποια άλλα θέματα. Με τα χαράς υποδέχομαι εξ την κυρία Μπάρμπαρα Βάιλερ, οποία είναι η συγγήτρια της Επιτροπής ασχολείται με την αναθεώρηση της ε, αναθεωρήσεως, με την εξέταση αναθεωρήσεως της οδηγίας για τις καθημερινές πληρωμές. Γίνεται πολύ σκληρή δουλειά σε επιτροπές. Η κυρία Μπάρμπαρα Βάιλερ προωθεί το χαρτοφυλάκιο στην Επιτροπή. Έκανε πάρα πολύ δουλειά ήδη. Ήδη διοργάνωσε μια δημόσια κρόαση με τους εμπλεκομένους και αφού ακούσουμε εσάς θα έχει το δύσκολο καθήκον να προτείνει τροπολογίες στην Επιτροπή να υποβληθούν στην Επιτροπή. Θα υπάρχουν δυνατότητες και για άλλες πολιτικές ομάδες να υποβάλουν τροπολογίες και μετά θα προτείνει συμβαστικές τροπολογίες και για την ψηφοφορία. Πολύ σημαντικό καθήκον και για κάθε εισηγητή. Στο κοινοβούλιο μας υπάρχουν και σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Βάιλερ είναι μέλος της ομάδας S&D, αλλά θα ακούσουμε και μέλη των άλλων πολιτικών ομάδων που είναι σκιώδεις εισηγητές και εκείνοι θα συμμετάσχουν στη συζήτηση και θα γίνει ανταλλαγή απόψεων θα ακουστούν οι απόψει απόψεις, οι δικέ σα. Με τα χαράς υποδέχομαι την κυρία Λιλιάνε Μπρίκμαν που είναι διευθύντρια τη Γενική Διευθύνσεω Επιχειρήσεων και βιομηχανία τη Ευρωπαϊκή Επίτροπή και βεβαίω όπω τα γνωρίζετε από τι συνθήκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα πρωτοβουλία. Έκαναν αυτή την πρόταση, μα την υπέβαλαν και τώρα δουλειά μα είναι να την ελέγξουμε και τη βελτιώσουμε. Θα δώσω τη δυνατότητα στην κυρία Μπρίκμαν να σχολιάσει αυτά που θα ακούσει από εσά αργότερα. Και κάτι άλλο να πω ότι από την αρχή που επεξεργαστήκαμε αυτή την πρόταση καλέσαμε την κυρία Μπρίκμα να μας παρουσιάσει την αξιολόγηση συνεπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόταση να μας δείξουν γιατί θεωρήσαν ότι χρειάζεται βελτίωση στους συγκεκριμένους τομείς μέσω αναλύσεως. Δεν είναι στο φάκελό σας σήμερα, αλλά για όσους δεν είδαν αυτό το έγγραφο ρίξτε το μια ματιά και ξέρω ότι αρκετοί από εσά ζητήσατε από τι εθνικέ σα αρχέ να εξετάσουν συγκεκριμένε αξιολογήσει συνεπιών ε, αυτής της πρότασης επί των οικονομιών σα. Τώρα, ποια είναι η ιδέα τη σημερινή ακροάσεω. Α, να καλωσορίσω με τα χαρά και υποψήφιο επίτροπο εσωτερική αγορά, τον κύριο Μισελ Μπαρνιέ, που ήρθε σήμερα ήρθε υπό την ιδιότητά του μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κόμμα, που είναι πλήρες και ενεργό μέλος της Επιτροπής. Με τα χαρά σας καλωσορίζουμε εδώ λοιπόν, πιθανότατα για τελευταία φορά σε αυτή την Επιτροπή, εκτός αν έρθετε και αύριο. Όμως είναι μεγάλη χαρά μας που είστε εδώ σήμερα. Έχουμε και μέλη των κρατών μελών, η Ισπανική Προεδρία εκπροσωπείται, διότι βεβαίως το Συμβούλιο επίσης ασχολείται με αυτή την πρόταση ταυτόχρονα Καλωσορίζω και αρκετούς εκπροσώπους άλλων κυβερνήσεων που παρίστανται και ίσως θα έχουν γνωστοποιήσει την παρουσία τους στους συναδέλφους. Μια-δύο παρατηρήσεις ακόμα. Ελπίζω να έχετε όλοι διερμηνία. Έχουμε διερμηνία σε 23 γλώσσες. Ελπίζω να ακούγεται καλά η διερμηνία. Αν χρειαζόστε βοήθεια, Έχουμε εδώ την ομάδα μας που μπορεί να σας βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα. Καλωσορίζω και πολλούς παρατηρητές που παρίστανται στην εδρίασή μας και θα, θα καλωσορίσω όλους ιδιαίτερος μια ομάδα μαθητών από την εκλογική περιφέρεια τη κυρία Βάιλερ, από ένα σχολείο τη εκλογική περιφερεια της κυρίας ήθελαν να παρακολουθήσουν τι κάνει. Και είναι πολύτιμο μέλο η κυρία Βάιλερ της εκλογικής περιφερειάς της κυρίας βαιλερ που ήθελα να παρακολουθησουν τι κανει και ειναι πολυτιμο μελο η κυρια βαιλερ της Επιτροπής μας. μακρηγορησα λιγο στην εισαγωγη μου αλλα ηθελα να δημιουργησω το σκηνικο οσον αφορα τη διαδικασια που θα ακολουθήσουμε, έχετε πρόγραμμα για τη συνεδρίαση. Θα χωρίσουμε σε δύο τμήματα τη συζήτηση. Υπάρχει ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για καθυστερημένε πληρωμέ στι δημόσιε αρχέ, κρατικέ αρχέ. Θέλω με αυτό να το εξετάσουμε συγκεκριμένα στο δεύτερο τμήμα τη συνεδριά σα, γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχόλιά σα. Οπότε θα χωρίσουμε τη συζήτηση σε δύο τμήματα και θα συμβάλλετε λοιπόν και στα δύο μέρη. Στο πρώτο τμήμα τη συνεδριά σα θα εξετάσουμε τι άλλε γενικέ πτυχέ των διατάξεων, συμβάσεων, κυρώσεις και άλλα γνωστά σας ζητήματα. Και η, η κυρία Βερνιού, η κυρία Μπερναντέν Βερνιού από τη Γαλλία θα προεδρεύσει αυτού του τμήματος και εγώ θα προεδρεύσω του δευτέρου τμήματος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα θέλαμε να ακούσουμε περισσότερο εσάς. Θα καλέσουμε λοιπόν όλους να μιλήσουν το πολύ για δύο λεπτά και θα έχουμε εδώ χρονόμετρο για κάθε τμήμα. Ελπίζω να μην είμαι πολύ περιοριστικό. Αν έχουμε περισσότερο χρόνο και λιγότερε παρεμβάσει, πάντα θα υπάρχει δυνατότητα δευτερολογία. Καλέσαμε του βουλευτέ να στείλουν. Ε, μια σελίδα το όνομά σας για να σας σημειώσουμε και έχουμε καταρτήσει κατάλογο ομιλητών. Θα καταρτήσουμε μάλλον. Αυτά για την ώρα. Καλώ την κυρία Μπάρμπαρα Βάιλερ καταρχά να θέσει το πλαίσιο και ο κ. Μπονασάρη από την Νομική Επιτροπή θα πει μερικά λόγια σχετικά με τι εργασίε εν λόγω Επιτροπή και ο κ. Ντεάντζελη τη Επιτροπή Βιομηχανία και Έρευνα και Ενέργεια θα μιλήσει. Διότι, τι γίνεται, εμεί είμαστε καθήλια αρμόδια Επιτροπή, αλλά η Νομική Επιτροπή και η Επιτροπή Βιομηχανία ενδιαφέρονται πραγματικά για το θέμα. Θα δώσω και σε αυτού δύο λεπτά στον καθένα για να θέσουν την προπτική τη επιτροπή του. Ε, θα είμαι πολύ αυστηρό στον φαρτοχρόνο. χρόνο. Η κυρία Βάιλερ έχει τετράλεπτο στη διαθεσή σα και μετά θα μπούμε στο βασικό τμήμα τη συζητήσεω. Ελπίζω τα πάντα να είναι ξεκάθαρα. Δίνω το λόγο τώρα λοιπόν στην κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου Καταρχήν να ε, καλωσορίσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και εγώ ήμουνα μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου μας και θυμάμαι ε, πόσο θέλαμε ήδη πριν τέσσερα χρόνια να ε, συμμετέχουμε στα όσα συνέβαιναν εκεί μακριά στις Βρυξέλλες. Ε, τότε δεν ήταν δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, τώρα όμως με τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι δυνατόν και ελπίζω να δράξετε και τη σημερινή ευκαιρία και τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στο μέλλον για να έχουμε αποτελεσματική νομοθέτηση. Η ιδέα της Κομισιόν Η πρωτοβουλία της Κομισιόν ε, για τις καθυστερήσεις των ε, πληρωμών, για τη βελτίωση των καθυστερήσεων των πληρωμών, ε, προέκυψε από, τις, από την πράξη, από τις καθυστερήσεις που υπάρχουν. Υπάρχει η επιθυμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια της Small Business Act να δουν βελτίωση των συνθήκων πληρωμής. Και επίσης η Κομισιόν με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στοχεύει στην ε, ε, εξάλληψη της γραφειοκρατίας. Οι καθυστερήσεις πληρωμών ε, δεν είναι δεν είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε πολύ ελαφριά. Δημιουργεί πραγματικό πρόβλημα. Και η σχετική πρόταση βοηθάει μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, λειτουργούν με αξιοπιστία. Υπάρχει η αρχική πρόταση της Κομισιόν από το 2000, η οποία τώρα αναδιατυπώνεται. Θα μπορούσε κανείς ε, να παρουσιάσει την επίκριση ότι θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει νωρίτερα, αλλά τώρα πραγματικά επήγει. Να πω επίσης καταρχήν ότι δεν έχω γράψει ακόμα την ε, έκθεσή μου. Περιμένω να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Πρόκειται δηλαδή για ακριβώς την σωστή στιγμή να ακουστεί η φωνή σας, να επηρεάσετε τις διαδικασίες. Το σημαντικότερο θέμα που ε, ε, θέλουμε να συζητήσουμε με εσά τους ε, βουλευτές είναι η εφαρμογή της οδηγίας. Ισχύει και για τις αρχές και για τους οικονομικούς φορείς. Προβλέπουμε όμως πιο αυστηρέ ποινέ για τις δημόσιες αρχές, διότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποτελούν υπόδειγμα και έχουν καλύτερες συνθήκες πλαίσιο, καλύτερη πρόσβαση σε πιστώσεις και διαφορετικό σχεδιασμό του προϋπολογισμού. Όπως και να έχει, δεν θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμός από τις δημόσιες ε, αρχές σε σχέση με τις ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Να σας πω ότι Όλοι βρήκαν υπερβολικά ψηλή την τιμή του 5% από όλε τι πλευρέ του Κοινοβουλίου ακούστηκε αυτό. Ε, θα πρέπει να βρούμε μια πιο λογική λύση με κάποια συγκεκριμένη κλίμακα. Επίσης ε, θα πρέπει να κλείσουμε κάποια παραθυράκια, κάποια κενά στη νομοθεσία, διότι δεν έχει νόημα η νομοθεσία που προβλέπει εξαιρέσεις για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση. Τέλος, αυτό που θέλουμε να εισάγουμε στην νομοθεσία είναι η κάλυψη και της Κομισιόν, η συμμετοχή και της Κομισιόν, όπως ε, αυτή ε, ισχύει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για ε, τις άλλες αρχές. Θέλουμε να εισάγουμε και το αγγλικό σύστημα της ε, προβολής των ε, καλών ε, περιπτώσεων. Αυτά είχα να πω εισαγωγικά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ Μπάρμπαρα. Θα έχεις τη δυνατότητα να συνοψίσεις το τέλος, οπότε θα ακούσουμε περισσότερο, περισσότερα πράγματα της Ο κ. Βαλτεσάρη έχει το λόγο για δύο λεπτά. Πρόεδρε, Χάρμπορ, η κυρία Βάιλερ, Επιτρέψτε μου πάνω απ' όλα να συγχαρώ, συγχαρώ για τη διοργάνωση αυτής της ε, ακροάσεως που ακολουθεί αυτή της 4ης Νοεμβρίου και εντάσσεται στην νομοθετική εργασία μιας αναθεωρήσεως οδηγίας που θέλει να ευνοήσει αναλογική ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς και απαιτεί όμως επαρκή διαβούλευση των εμπλεκομένων μέρων. Χαιρετίζω βεβαίως τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η νέα πρόταση σαν στόχο έχει βασικό να βελτιώσει και να παγιώσει την εφαρμογή της ε, ε, οδηγίας 2035. Το νέο κείμενο κάνει διάκριση θεμελιώδη μεταξύ επιχειρήσεων που οφείλουν, έναντι των οποίων η οδηγία προβλέπει δυνητικής ευχέρειας μέτρα διορθωτικά και επίσης και δημόσια δίκηση που χρωστάει χρήματα, όπου εκεί υπάρχουν δυνατότητες προσφυγής που είναι αυτόματα μέσα ε, και μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιηθούν. Λοιπόν, ε, είναι πιο αυστηρή η πρόταση αυτή εν συγκρίση έναντι της δημόσιας διοίκησης. Πρέπει να δούμε τι κάνει η μελέτη ε, συνεπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έδειξε αυτή η μελέτη όμως ότι όσον αφορά τις πληρωμές υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή η αξιολόγηση συνεπιών. Γιατί έγινε αυτή η επιλογή ότι οι δημόσιες αγορές των κατομελών το 2006 ήταν πάνω από 1.943 δις ευρώ και επηρέαζαν ουσιαστικά την ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με αυτό, βασιζόμενο σε αυτό, θα ήθελα να περιοριστώ σε αυτό που πιστεύω ότι είναι ένα από του βασικού ε, στόχου τη ακροάσεω αυτή. Χωρί να επισέλθω στην ουσία τη προτάσεω, που μπορούμε να συζητήσουμε ενδελεχέστερα αργότερα. Πιστεύω ότι η σημερινή ακρόαση είναι θεμελιώδη σημασία για να επισημάνουμε κάτι Δηλαδή, ποια πρόταση πρέπει να ακολουθήσουμε για την ε, νομοθεσία μα και για την πρόταση. Θέλουμε ισορροπημένο τελικό κείμενο που να μπορεί να είναι ένα κίνητρο και να μην καταδικάζει τι χώρε που έχουν πρόβλημα. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι χρειάζεται να πλαισιώσουμε ελιστικό τρόπο την όλη προβληματική και να δράσουμε νομοθετικό πώ προ σκοπών επίτευξη στέρεη βάσεω για αρμονική ανάπτυξη εσωτερική αγορά και σταθμίζοντα τις δεσμεύσει του Μάστρικ από μια πλευρά και από την άλλη τι υποχρεώσει και τι δυνατότητε που έχουν στο πλαίσιο του προπολογισμού του στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που εστιαστήκατε στα θέματα που αφορούν περισσότερο την Επιτροπή σας. Και ο κύριος Ντι Άντζελης έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ ο πρόεδρε Χάρμπορ, ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Βάιλερ. Επικροτώ αυτή την πρωτοβουλία, πραγματικά πολύ χρήσιμη διότι τώρα μπαίνουμε στην φάση τη σημαντικότερη, την πιο σημαντική θα έλεγα, πάνω σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι ιδιαίτερα αισθητό στην Ευρώπη. Χαιρετίζω όλους τους εθνικούς ε, βουλευτές. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει πολύ, βαρύνει πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βαρύνει πάνω απ' όλα τις επιχειρήσεις σε μια στιγμή μεγάλης κρίσεως, διεθνούς κρίσεως, που πλήττει τόσες επιχειρήσεις, τόσες οικογένειες, πάνω απ' όλα τόσους εργαζομένους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως λέει και η συγγήτρια, να δούμε ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή. Είναι, θέλουμε μια οδηγία που θα βρίσκει λύσεις, κυρίως αυτό. Να μπορεί να βρει απάντηση, να δώσει απάντηση σε ένα πρόβλημα που βαρύνει και κάνει να σφιχτούν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα ερχόμενοι στο θέματα που αφορούν περισσότερο την οδηγία. Κάποια ζητήματα να θέσω. Πρώτα απ' όλα, το επέκταση του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας. Αυτό είναι ένα θέμα συζητήσεως. Και ο χρονικός συντονισμός όσον αφορά τις διαγραφές, τα, περίο, τα περιθώρια, να μειωθούν τα περιθώρια ε, παρεκκλήσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μειωθεί το περιθώριο παρεκκλήσεων και εξαιρέσεων, το δικαίωμα των επιχειρήσεων να ενημερώνονται. Όσον αφορά αυτό το θέμα λοιπόν, να γίνει μια εκστρατεία ενημέρωσης πολύ διεξοδική και αποτελεσματική. Αυτά είναι κάποια τα σημεία, κάποια από τα χρήσιμα σημεία προς συζήτηση σε αυτό το διάλογο. Αναμφισβήτητα μετά όταν θα μπούμε στην ουσία και θα αρχίσουμε στις 4 του μήνου στην Επιτροπή Ήτρε το, της του θέματος να μπορέσουμε πιο άμεσα, πιο αποτελεσματικά να εμβαθύνουμε και να δώσουμε απάντηση για μια οδηγία που θα δίνει απαντήσεις σε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να σβήσετε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Καλώς. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για τις αφέστατες εισαγωγές αυτές. Θα δώσω τώρα την Προεδρία στην Αντιπρόεδρό μας την κυρία Βανιέ, η οποία θα διευθύνει το πρώτο ήμιση της συζητήσεως οπότε έχει το λόγο Μπερνάντετ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Το ζητήσαμε, ελπίζαμε να έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και την έχουμε. Και έτσι μπορούμε τώρα όλοι μαζί 27 χώρες να συνεργαστούμε μαζί με εσά ώστε να έχουμε μια εσωτερική αγορά λιγότερο κατακαιρματισμένη. Από αυτό θα επωφεληθεί ο κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση. Θα είμαι σύντομη. Η οδηγία αυτή κάνει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Στο πρώτο τμήμα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έχετε λοιπόν δύο λεπτά ο καθένας από εσά και θα σας ζητήσω να τηρήσετε το χρόνο σας. Έτσι θα μετράμε το χρόνο. Θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ζωζέ Ντιρμπέιρου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, αλλά εγώ θέλω το λόγο στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης, παρακαλώ. Καλώς. Τότε δεν είχα το σωστό σημείωμα μπροστά μου. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Ιρλανδία. Ο κύριος Μικελ Ράιν έχει το λόγο. Μάικλ Ράιν. Κι εγώ για το δεύτερο μέρος ε, έχω γραφτεί. Στο δεύτερο τμήμα θέλω να πάρω το λόγο. Α, δεν πάμε καλά, λέει η κυρία Βερνιό. Τώρα, Κωνσταντ Λίνκ. Ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη και τα γραφά μου και δεν άκουσα το όνομά μου αμέσω. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, κυρία Ισηγήτρια, σα χαιρετίζω θερμά όλου και όλε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να πάρω το λόγο εδώ, σε αυτό το τμήμα μια που η τροποποίηση της οδηγίας, στην οποία αναφερόμαστε σήμερα, είναι κάτι που περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κυρίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Διότι ακριβώς οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που ενδιαφέρονται όλος ιδιαίτερος για την άμεση εφαρμογή της οδηγίας αυτής, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε κατά πόση οδηγία ασχολείται μόνο με τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις σχέσεις τους. Στη χώρα μου, το θέμα των καθυστερήσεων πληρωμών δεν έχει να κάνει μόνο με συναλλαγές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με τον δημόσιο τομέα, αλλά υπάρχουν τέτοια προβλήματα και στις σχέσεις των επιχειρήσεων των ιδιωτικών μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί τις λειτουργίες στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πολύ συχνά τονίζουν ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών από πλευράς του δημοσίου τους δημιουργεί ζημιά, γιατί πρόκειται για σημαντικά ποσά πολλές φορές. Αν λοιπόν η πληρωμή δεν γίνεται έγκαιρα, τότε κινδυνεύει η ρευστότητα των επιχειρήσεων αυτών. Είναι τέτοια τα ποσά που οι επιχειρήσεις δεν μπορούν από την άλλη μεριά να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε άλλες επιχειρήσεις, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν που είναι επίση σημαντικό είναι οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων να συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία. Οι ίδιες επιχειρήσεις λένε ότι κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε τη λειτουργία τους και θα τις έκανε πιο αποτελεσματικές στη λειτουργία τους. Είναι κάτι που έχουν υπογραμμίσει εκπρόσωποι μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως επίσης και το ότι χρειάζεται μία διάταξη η οποία να εμποδίζει, για παράδειγμα, τους μεγάλους διανομής να επιβάλλουν στους μικρούς προμηθευτές προθεσμίες πληρωμών που να ξεπερνάνε τις εκατομέρες σε μερικές περιπτώσεις. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, εδώ πρόκειται και για το δικαίωμα ίσπραξης των διοικητικών δαπανών. Ένας από τους λόγους των προσφυγών που έχουμε είναι ότι υπάρχουν έξοδα για την ίσπραξη που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε καλό θα ήταν να υπάρχει και μια τέτοια διάταξη θα βοηθούσε πάρα πολύ τις επιχειρήσεις εφόσον συμπεριλαμβάνονταν κάτι τέτοιο στην οδηγία. Αυτό θα βοηθούσε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να εισπράττουν τα χρήματά τους. Και τέλος, κάτι για το οποίο επιμένω και προς τους συναδέρφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση, ενημέρωση για το ότι μπορεί κανείς να προσφύγει στην οδηγία αυτή. Ξέρω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, συγγνώμη, λέει Μιλήτρια. Καλώς. Να τηρείτε το χρόνο σας, τα δύο λεπτά. Δεν έκοψα τη συνάδελφο, αλλά είναι σημαντικό να τηρούμε το χρόνο μας, γιατί έχουμε εδώ τα εθνικά κοινοβούλια, δεν τα έχουμε εδώ κάθε μέρα. Οπότε καλό είναι να του δοθεί ευκαιρία να μιλήσουν. Η κυρία Βαχόκ τώρα. Για το πρώτο τμήμα θέλει να μιλήσει ή για το δεύτερο, για να ξέρουμε. Παρακαλώ. Α, εντάξει. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Εκ μέρους της Γερμανίας. Κύρια Πρόεδρε, κύρια εισηγήτρια, ναι, ευχαρίστω θα μιλήσω στο, δε... πρώτο μέρος της συζήτησης, αλλά αν μου δώσετε και ένα λεπτό ε, στο δεύτερο μέρος για να μιλήσω για τη διαφορά ανάμεσα στις ε, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, αυτό θα ήταν πολύ καλό. Ε, έρχομαι από το ε, Γερμανικό Bundestag, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και χαίρομαι ιδιαίτερα με αυτό που έχουμε τώρα στη συνθήκη τη Λισαβόνα, την ε, στενότερη συνεργασία δηλαδή με τα εθνικά κοινοβούλια. Πολύ ευχαρίστω θα συμμετάσχουμε στο μέλλον σε περισσότερες συζητήσεις ε, για να επηρεάσουμε τι διαδικασίες. Ως εκπρόσωπο Εθνικού Κοινοβουλίου στην οδηγία αυτή με ενδιαφέρει το κατά πόσο είναι συμβατή με την εθνική μας νομοθεσία. Αυτό βέβαια είναι αυτονόητο, αλλά απλά ήθελα να το αναφέρω και ως ε, Γερμανίδα πολιτικός θέλω να τονίσω ότι δεν πρέπει να το επίπεδο προστασίας να είναι ε, χαμηλότερο με την οδηγία. Επίσης, ε, στο άρθρο 5 έχουμε το 5% τα αποζημίωσης. Η κυρία Συγήτρια ήδη είπε ότι πολλοί θεωρούν ότι το 5% αυτό είναι υπερβολικά ψηλό. Θα χαρούμε αν ε, επιλεγεί ένα χαμηλότερο ποσοστό ωστόσο θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητο αυτό το μέτρο αποζημίωσης στην οδηγία αυτή, διότι υπάρχουν άλλα μέτρα αποζημίωσης. Ε, θα παρακαλούσαμε λοιπόν ε, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την ε, Κομισιόν να διαγράψουν τελείως το ποσοστό αυτό της αποζημίωσης και να θεωρήσουν ότι αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 αρκούν ε, για να ε, δημιουργηθεί μια καλύτερη ε, συμπεριφορά των οφειλετών. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Je pense que vous avez... Ευχαριστώ. Τηρήσατε το χρόνο σας, οπότε πρόεδρε Ίσως το δεύτερο γύρο να μπορεί να έχει ένα λεπτό παραπάνω. Τώρα, το λόγο έχει η πολωνική γερουσία, ο κ. Σούλεβιτς. Δεν ξέρω αν πρόφερα καλά το όνομά σας, τα πολωνέζικά μου δεν είναι πολύ καλά. Ευχαριστώ. Πολύ καλά προφέρατε το όνομά μου. Σας ε, χαιρετίζω όλους εκ μέρους της Πολωνικής Δημοκρατίας και του Πολωνικού Κοινοβουλίου. Το θέμα των πληρωμών τώρα, των καθυστερήσεων πληρωμών, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που έχει άμεση σχέση με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Μπορεί να μην φαίνεται αυτό πολύ εύκολα, αλλά είναι γεγονός ότι επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Όλα αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με την κρίση, έχουν να κάνουν με την οικονομική συγκυρία και σε κάθε εποχή κρίσης οι πληρωμές καθυστερούν ακόμα πιο πολύ. Αυτό είναι κάτι που έχει ιδιαίτερα να κάνει με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό πιστεύω στη συζήτησή μας ότι πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώς σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εκείνες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα κάθε φορά που πρέπει να εισπράξουν χρωστούμενα, οφειλές. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Το 5% πιστεύω και εγώ ότι είναι κάπως υπερβολικό. Θα έπρεπε σταδιακά να υπάρχουν ε, οι κυρώσεις με διάφορες κλίμακες και να μην έχουμε τις ίδιες κυρώσεις για κάποιον που έχει καθυστερήσει μια μέρα και τις ίδιες με κάποιον άλλον ο οποίος έχει καθυστερήσει δεκαήμερα ολόκληρα. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε και να το τονίσουμε, γιατί μικρές και μεσές επιχειρήσεις φοβούνται ότι όταν προσπαθούν να εισπράξουν οφειλές, αυτό το οποίο θα συμβεί είναι ότι θα χάσουν τους πελάτες τους. Αυτό είναι ο μεγάλος φόβος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε ότι άμα χάσουν τους πελάτες τους, για αυτές τις επιχειρήσεις είναι πολύ σοβαρό και οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερε καθυστερήσει. Είναι ένα φαύλο κύκλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο τώρα στου και ηγητή και του φιλελευθέρου, τον κύριο Γιώργεν, Γιώργεν Κάτσμαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο πράγματα θα ήθελα να αναφέρω στην ε, εισαγωγική παρέμβαση αναφέρθηκε το θέμα ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις συχνά εποφελούνται από το σύστημα, γι' αυτό θα βοηθούσε τις μικρές επιχειρήσεις να θεσπιστεί μια προθεσμία μέγιστη για τις πληρωμές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 60 μέρες για παράδειγμα. Θα ήθελα να σας θυμίσω επίσης όσον αφορά την αποζημίωση 5% ότι όταν μιλάμε για 100 ευρώ μιλάμε για 5 ευρώ, για, ε, αν μιλάμε για 1000 ευρώ το 5% είναι 50 ευρώ, αν μιλάμε 10, για 10.000 ευρώ μιλάμε για 500 ευρώ. Αν συνεχίσουμε ε, αν μιλάμε για ένα εκατομμύριο, μιλάμε για 50... Ε, ε, για 50.000 ευρώ. Στόχος εδώ πέρα ποιος είναι. Είναι να γίνονται οι πληρωμές εγκαίρως, διότι σε κοινοτικό επίπεδο διαπιστώνουμε ότι ακόμα και για, μικρότερες, ε, για μικρότερα ποσά πληρώνονται ποινές. Τα αγγλικά νοσοκομεία λένε ότι όλα πάνε πολύ καλά, διότι οι πληρωμές ε, γίνονται ε, πρόθεσμα στο 90% των περιπτώσεων, αλλά και για το υπόλοιπο 10% θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Φυσικά, στο γερμανικό σύστημα είναι ε, ξένο στοιχείο το να εισάγεται αποζημίωση για καθυστέρηση πληρωμών, διότι αυτό γίνεται με την ίσπραξη τόκων. Αυτά. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στο Λόρδο Μπάουνες. Uh, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή την ακρόαση. Η Επιτροπή της Βουλής των Λόρδων, που, της οποίας προεδρεύω, εξετάζει το θέμα και να πω ότι πραγματικά έχουμε απογοητευτεί τα μάλα με την αξιολόγηση συνεπειών που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε υποθέσεις σχετικά με την ανάγκη για θέσπιση νομοθεσίας χωρίς να υπάρξει διαβούλευση με πολλούς. Τούτου λεχθέντος, βεβαίως ως Επιτροπή δεχόμαστε ότι η καθυστέρηση πληρωμών είναι πρόβλημα στα κράτη-μέλη και θέλουμε να αλλάξει η νοοτροπία και να καταβάλλονται άμεσα πληρωμές και έχει ιδιαίτερε συνέπειε για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις για λόγους που αναφέρθηκαν οι μικρές επιχειρήσεις είναι πιο πιθανόν να απόσχουν από την πίεση για την καταβολή οφειλωμένων πληρωμών λόγω εμπορικών σχέσεων με τους μεγαλύτερους εταίρους τους. Κρίμα που η πρόταση δεν έχει σαν στόχο πιο συγκεκριμένα τις μικρές επιχειρήσεις. Όσον αφορά το έγγραφο Τσιγήτρια, συμμεριζόμαστε την ανησυχία που εκφράζεται ότι η καταβολή αποζημίωση πέρα του τόκου για 1%, 1% για χρέη πάνω από 10.000 ευρώ, αυτό είναι κάτι εντελώ δυσανάλογο, είναι κάτι ανάλογο με κύρωση, δεν θα πρέπει να περιγράφεται ω αποζημίωση. Θέλουμε λογική καταβολή πληρωμών που σχετίζονται με το εμπλεκόμενο κόστος και μπορεί να ζητηθεί καταβολή συμπληρωματικού κόστους που θα, αντι... θα αντικατοπτρίζει το πραγματικό συμπληρωματικό κόστος που προκύπτει. Λοιπόν, χρειάζεται συζήτηση με τις επιχειρήσεις γι' αυτό. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα ποσά μπορεί να ανακτηθούν ως αποτέλεσμα δικαιώματος, αλλά και πάλι θα πρέπει να προσφύγουν οι μικρές επιχειρήσεις εάν δεν πληρωθούν. Επιτρέψτε μου να μιλήσω αργότερα, κυρία Πρόεδρε, στο θέμα αυτό για την πρόταση για το δημόσιο τομέα. Ήσασταν ακριβέστατος. Σας ευχαριστώ όσον αφορά το χρόνο. Θα δώσω το λόγο στην Καταλωνία, στον κύριο Τζόρντι Βιλατζουάνα, για τη Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μας δίνει την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας εδώ. Συμφωνούμε απόλυτα για την ε, ανάγκη που υπάρχει να ρυθμιστεί η κατάσταση, δεδομένη της τόσο δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουν ε, πολλές ε, χώρες, οικονομικά δύσκολοι. Υπάρχουν δυσκολίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα. Στην Ισπανία έχουμε ε, μια προσπάθεια για ένα νέο νόμο προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και οι προτάσεις της Κομισιόν. Προτερότητά μας, όπως και της Κομισιόν, είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και ένα άλλο στοιχείο κλειδί για την Ισπανία, πολύ σημαντικό, είναι οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες, οι αυτόνομοι. πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο 60 ημερών και να φροντίσουμε να εφαρμόζεται το μέτρο των 60 ημερών. Στις περιπτώσεις που δεν τηρείται, να φροντίσουμε για το ποια θα είναι η κύρωση, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη με την οφειλή, ανάλογη με το ποσό της οφειλής. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από τις κυρώσεις. Εμείς λέμε ότι μπορεί να φτάνει και το 15%. Αλλά Ξέρω ότι είναι ένα στοιχείο κλειδί εδώ. Και το θέμα των τόκων και ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια αύξηση της τάξης του 50% για να υπάρχει μια σαφή σκήρωση για αυτούς που δεν τηρούν τις προθεσμίες πληρωμής. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να προστατεύσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως επίσης και τους αυτόνομους, ότι 60 μέρες είναι μια πρώτη προθεσμία καθοριστική, στη χώρα μου έχουμε και παραπάνω, και για το δημόσιο τομέα, όπως είπε και ο συνάδελφος πριν, θα επανέλθουμε στο δεύτερο τμήμα. Και εκεί πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε όριο τις 30 ημέρες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα, Χάιντερ Χούλε, σκιώδης για τους πρασίνους. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Μια πολύ μικρή παρατήρηση θέλω να κάνω και για τον ε, δημόσιο τομέα, διότι μάλλον δεν θα μου δώσετε το λόγο. Εγώ ε, πιστεύω στην ίση μεταχείριση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, διότι πιστεύω ότι άμα θέλουμε να βελτιώσουμε την οτροπία πληρωμών στην Ευρώπη, και αυτό είναι ο στόχο τη ε, οδηγία αυτή, δεν έχει νόημα να δημιουργούμε νέε ανισότητε και στρεβλώσει στην αγορά. Και αυτό θα συμβεί εάν μεταχειριζόμαστε διαφορετικά τον ιδιωτικό από τον δημόσιο τομέα. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τα ιδιωτικά νοσοκομεία σε σχέση με τα δημόσια. Αυτό δεν ε, θα βελτιώσει την ε, κατάσταση. Πιστεύω επίσης ότι για να βελτιώσουμε την κατάσταση θα πρέπει να έχουμε και θετικά κίνητρα, όχι μόνο αρνητικά, όχι μόνο ποινές δηλαδή, κυρώσεις. Και το naming and shaming, το να προβάλλουμε τα κακά παραδείγματα ε, δεν γίνεται σε όλες τις χώρες, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε και θετικά κίνητρα και αυτό το έχει παραμελήσει η Κομισιόν. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να εισάγουμε τις 30 μέρες προθεσμία χωρίς εξαιρέσεις. Ε, θα πρέπει να είναι οριστική, ε, οριστικό το τιμολόγιο. Επίσης, ε, συμμερίζομαι τη θέση πολλών προλαλισσάντων ότι είναι υπερβολικό να ε, ζητάμε αποζημίωση 5% ήδη από την πρώτη μέρα καθυστέρησης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε πιο σοφά, να σκεφτούμε πιο μακροπρόθεσμα και γι' αυτό πρότασή μου θα είναι αυτή που ακούστηκε επίσης. Στους στόχους υπερημερίας να προσθέσουμε ένα ή 2% με ποινή 5% πιστεύω ότι ε, δίνουμε χώρο και στους κερδοσκόπους που θα θέλουν να βάλουν στην τσέπη τους τα 5% αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα στο Πολωνικό Κοινοβούλιο Λόγος. Πάουελ Πόνσι Σίλστ, ενδεχομένως, συγγνώμη για την προφορά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε αυτό το πρώτο τμήμα της συζητήσεώς μας θα ήθελα να αφαιθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο, σίγουρα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση όσον αφορά την εναρμόνιση του προβλήματος της καθυστερήσεως πληρωμών στα διάφορα κράτη-μέλη. Απ' την άλλη, πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι οι προσδοκίες μας να λύσει όλα τα προβλήματα η οδηγία είναι κάτι μάταιο, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαφορα κάτι κράτη-μέλη. Αυτές οι καθυστέρησεις πληρωμών επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σε, σε βασικό ποσοστό και λιγότερο τη βιωσιμότητα των δημοσίων φορέων. Στο Πολωνικό Κοινοβούλιο δεν έχουμε σήμερα δεν συζητούμε το πρόβλημα καθιστής πληρωμών του δημόσιου τομέα έναντι των ιδιωτών. Το πρόβλημα που μας αφορά κυρίως είναι το, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στον φάση καθυστέρησης πληρωμών. Επιμένω πάνω σε αυτό. Αυτή είναι η οδηγία που μου έδωσε η Οικονομική Επιτροπή του Πολωνικού Κοινοβουλίου. Άλλα σχόλιά μου αφορούν τα άρθρα της νέας οδηγίας, κυρίως το 4, το άρθρο 4, οι άγνωστες διατάξεις εμπεριέχονται, άγνωστες διατάξεις για τον πολωνικό νόμο, οι αποζημιώσεις εξαρτώνται πάνω απ' όλα από τη βλάβη, από τη ζημιά. Και αυτή η αποζημίωση μοιάζει με συμβατική κύρωση. Στο άρθρο 7 Κατά την άποψή μας, χρειάζεται συμπλήρωση. Χρειάζεται κάποια διάταξη που θα επέμενε επί της υποχρεώσεως που υπέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη να δίνει πληροφορίες που θα επιτρέπει στα νομικά συστήματα και στα θεσμικά όργανα των κρατών μελών να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία όσον αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών και, τα, και τους τόκους που θα πρέπει να καταβάλλονται για καθυστερήσεις οφειλωμένων πληρωμών στα εμπορικά ζητήματα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Το Ιταλικό Κοινοβούλιο, ο κ. Τζοβάνι Φάβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ απηχώ τη συζήτηση που ξεκίνησε ήδη στην αρμόδια επιτροπή στη, στο Ιταλικό Κοινοβούλιο και εκεί έγιναν, πρότεινα και εγώ κάποιο ψήφισμα τις προάλλες που ακολουθεί την κατεύθυνση που ήθελαν πολλοί από προλαλήσαντες. Πιστεύουμε ότι αυτή η διάκριση που γίνεται με, για την εφαρμογή, διάκριση δική μεταξύ δημόσιας διοίκησης και επιχειρήσεων, αυτή η διάκριση δημιουργεί διαφοροποίηση όσον αφορά την αγορά, κάτι απαράδεκτο. Πέραν από αυτό, ε, στη χώρα μας αντιμετωπίζει το εξή φαινόμενο. Δύσκολη δυσχέρεια που δημιουργεί το σύστημα των πληρωμών στις μεγάλες δομές ε, διανομής που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις. και εν συγκρίση μάλιστα με έναντι των δημοσίων δικήσεων. Πιστεύουμε και εξεκολουθούμε να πιστεύουμε ότι έχει προτεραιότητα αυτή η οδηγία κατά κάποιο τρόπο να κάνει να συμπέσουν, να συγκλίνουν τα, τα συμφέροντα των δύο πλευρών που διαχωρίζονται σε αυτή τη φάση. Και δεν μπορούμε παρά να αναφέρουμε κάποιες διαφορές που θεωρούμε διαφοροποίησεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν στους δύο τομείς. Στον ιδιωτικό τομέα, το, ο χρονικός συντονισμός ε, πληρωμών πρέπει να ποικίλει μεταξύ 60 και 90 ημερών. Πρέπει στη δική μας ένωμη τάξη χρησιμοποιήθηκε. Ποτέ δεν το αντιληφθήκαμε διαφορετικά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών στον αφορά τις επιχειρήσεις, ούτε επιχειρήσεις το βλέπουν διαφορετικά. Πρέπει τελικά θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι χρόνοι πληρωμών, να αλλάξει η νοοτροπία. Είναι κάτι που ταλαιπωρεί όχι μόνο τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, ε, σχέση με τη δημόσια ε, διοίκηση, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των διαφόρων μεγάλων δικτύων ε, διανομής, που δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο σκιώδη, τον κύριο Έντουαρτ Σοσούσνικ, δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, μπορεί να εξοικονομήσω κάποιο χρόνο υπενθυμίζοντας τους βασικούς δισταγμούς που είχαμε κατά διάρκεια των συζητήσεων όταν συζητήθηκε στην Επιτροπή ΙΜΚΟ στις 28 Σεπτεμβρίου και στην πρώτη συνάντηση της Επιτροπής αυτής είπα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή η πρόταση είναι πολύ δυσνόητη καταρχάς ε, εμπεριέχει πτυχές που ευνοούν τη διαφθορά. Αν κάποιος υπάλληλο αποφασίσει να κοιμηθεί Φερρυπίν, όσον αφορά μια σύμβαση που αφορά εκατομμύρια ε, ευρώ, αν δεν προσέξει, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα και να ευνοηθούν κάποια συμβαλόμενα μέρη της, ε, του δημόσιου τομέα. Κάποιοι που προμηθεύουν επιχειρήσεις με αγαθά ή τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και η αξιολόγηση συνεπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι απόλυτα πιστική. Παρόλο που εμπεριέχονται και κάποια θετικά στοιχεία. Καμιά φορά υπάρχουν μεγάλε καθυστερήσει σε διάφορα κράτη-μέλη. Επί εκατοντάδε ημέρε υπάρχουν καθυστερήσει. Ενώ στη Γερμανία και στη Τσεχία, Φερρυπίν, δεν υπάρχουν τέτοιου είδου μεγάλα προβλήματα. Τελικά θα βρούμε συμφωνία αν σεβαστούμε κάτι βασικό. Όλες οι πολιτικές ομάδες. Δηλαδή να είναι ισότιμες οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Λοιπόν, Σα ευχαριστώ που σέβεστε το χρόνο αγορευσή. Είσαστε ακόμα, μιλάτε ακόμα και λιγότερο. Νομίζω ότι δεν θα απογοητευτούμε το απόγευμα, θα μπορούσαμε να ξαναδώσουμε το λόγο σε όσου επιθυμήσουν να δευτερολογήσουν. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο για τα εθνικά κοινοβούλια, η Ελλάδα και η Ισπανία. Να δώσω το λόγο στον κύριο Χρήστο Πρωτοπαπά για την Ελλάδα, για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο. το μικρόφωνο σας. Ακούγεται τώρα, ναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω μόνο για το κομμάτι που αφορά το ιδιωτικό τομέα και θα παρακαλούσα να μου ξαναδώσετε το λόγο για το δημόσιο εν συνεχεία στο δεύτερο γύρο. Ε, είναι σαφές ότι για το κομμάτι που αφορά τον ιδιωτικό τομέα η οδηγία μπορεί να δράσει θετικά. Ούτω ή άλλω, μα ενδιαφέρει να υπάρχει ανάπτυξη και τόνωση τη αγορά σε σημερινέ συνθήκε. Είναι σαφέ ότι η αλλω μας ενδιαφερει να υπαρχει αναπτυξη αυτή σημερινέ συνθηκες ειναι σαφες οτι στηρίζεται και στο Small Business Act του 2008. Μας ενδιαφέρει να ε- ε- ε- βελτιωθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και να βελτιωθεί η ρευστότητά τους. Και είναι σαφές ότι η καθυστέρηση πληρωμής συνιστά μεταφορά ρευστότητας από τον πιστωτή στον οφηλέτη. Ε, άρα είναι σαφές ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα. Θεωρώ ότι με την προσπάθεια που γίνεται βελτιώνονται τα μέτρα που προβλέπονται από παλαιότερα. Ε, θα πρέπει βεβαίω να εξηγήσουμε με ποιο κριτήριο μπαίνει αυτό το 1% για τις περιπτώσεις καθυστερήσεων μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σε κάθε όμως περίπτωση, και το λέω από τώρα, το 5% που έχει να κάνει με την ε, διαφορά για τις περιπτώσεις καθυστερήσεων του δημοσίου με επιχειρήσει στι οποίε οφείλει χρήματα είναι εξόχω δυσβάστακτο και αρνητικό, όχι απλά υπερβολικό, εξόχω δυσβάστακτο και αρνητικό και πρέπει να αλλάξει. Συμφωνούμε λοιπόν επί της αρχής για την προσπάθεια. Χρειάζεται να πάρουμε κάποια μέτρα για να βελτιώσουμε τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να τονώσουμε τι αγορέ. Το μέτρο αυτό λειτουργεί σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει όμω να αποφύγουμε τι υπερβολέ και το 5% είναι μια υπερβολή που μπορεί να δημιουργήσει παρά να λύσει προβλήματα ειδικότερα για το δημόσιο τομέα, θα τα πω στη δεύτερη παρέμβασή μου. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Φέλιξ Λαρόζα Πικέ για το Ισπανικό Κοινόβουλιο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Κομισιόν, προκειμένου να έχουμε συνομιλία όλα τα εθνικά κοινοβούλια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Και εποφερούμε από την ευκαιρία αυτή, να πούμε και και τελευταίο ομιλητή σε αυτό το πρώτο μέρος, για να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην εισηγήτρια, προκειμένου να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Συγχαρητήρια και σε όλε τι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου που βοηθάνε. Πρέπει να καταλήξει θετικά αυτή η υπόθεση, γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς εξαρτιόμαστε από αυτό που θα αποφασίσετε εσείς. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ στο Ισπανικό Κοινοβούλιο και όπως είπε και ο συνάδελφος, συζητιούνται διάφορες πρωτοβουλίες στην Ισπανία για να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα αυτά που έχουν να κάνουν με τις καθυστερημένες πληρωμές. Συμφωνώ με πολλές από τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν εδώ. Συμφωνώ επίσης και με αυτά που είπε ο σκιώδης εισηγητής, ότι δηλαδή πρόκειται για καταστάσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις δυστυχώς σε ορισμένες χώρες πλήττονται περισσότερο οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις από ό,τι σε άλλες είναι θέματα που έχουν να κάνουν με την οτροπία που ισχύει στην κάθε χώρα. Ελπίζουμε, πας περιπτώσει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, καταλήξει σε μια σύγχρονη πρωτοβουλία η οποία στην πράξη να μπορεί να βοηθήσει να πετύχουμε δηλαδή το στίχο μας που είναι να πληρώνονται οι οφειλές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τις λιγότερες δυνατόν καθυστερήσεις προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να πληρώνονται όσο γίνεται λιγότερο οι τόκοι υπερημερίας. Βέβαια, πονάει λιγάκι το γεγονός ότι οι νομοθέτες πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ό,τι ότι νόμο εγκρίναμε παλιότερα δεν βοήθησε στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και θα ολοκληρώσω με το εξή. Μην κοιτάμε μόνο τις προθεσμίες πληρωμών, όταν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των ε, διαφόρων πλευρών, όταν για παράδειγμα ο διατροφικός τομέας συμφωνεί για κάποιες προϋποθέσεις, για προθεσμίες πληρωμές, αυτό αποτελεί μέρος ενός περιεχομένου, ενός συνόλου διαπραγματεύσεων όπου συζητιέται για παράδειγμα και σε ποιο ράφι στο σούπερ μάρκετ θα μπει το συγκεκριμένο τρόφιμο. Αυτό θέλω να σας ε, το πω για να το έχετε υπόψη σας όλοι. Όπως και να έχουν τα πράγματα πάντως, θα ήθελα να σας ζητήσω να μη σκεφτόμαστε μόνο τις κυρώσεις, μόνο τις ποινές. Ακούστηκε ότι πρέπει να δούμε λίγο και πώς θα προωθήσουμε ένα κώδικα διοντολογίας. Είναι σημαντικό επίσης για το θέμα της ε, εκπροσώπησης να το λάβουμε υπόψη μας. Ποιος εκπροσωπεί ποιον. Έπειτα υπάρχουν και άλλες εγγύσεις που νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στα πλαίσια αυτής της οδηγίας. Συγγνώμη αν ε, καθυστέρησα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Τώρα, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιώδης συζητητής, ο κύριος Δεγιόν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι Πολύ σωστά, οι περισσότεροι που πήραν εδώ το λόγο τόνισαν το θέμα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Όντως, και εμείς στην Ολλανδία το έχουμε ακούσει από τις μικρές επιχειρήσεις το πρόβλημα πολλές φορές, πόσο πιέζονται Στην μεταλλουργία επίσης οι προμηθευτές λένε ότι δεν τους είναι εύκολες οι προθεσμίες τις οποίες συζητάμε. Οι καθυστερήσεις φτάνουν ε, ένα εξάμεινο πολλές φορές. Αναγκάζονται όμως να τα δεχτούν όλα αυτά. Η Επιτροπή με την έκθεση αντικτύπου, με τη μελέτη αντικτύπου, προσπαθεί να δει πώς έχουν τα πράγματα στην αγορά και να ξέρει προς τα πού πρέπει να προσανατολιστεί. Πάντω δεν είναι δυνατόν πίσω από την ελευθερία της κάθε σύμβαση να κρυβόμαστε και έτσι τελικά να ζημιώνονται οι επιχειρήσεις. Αν είσαι μια μικρή επιχείρηση δεν έχει πραγματικά ελευθερία να διαπραγματευτείς όπως θα περίμενε κανείς. Οπότε θα έλεγα να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στις επιχειρήσει τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο τομέα. Αυτό σίγουρα. Αλλά Οι 30 μέρες θα πρέπει να είναι ο κανόνας και από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε για μικρές επιχειρήσεις που έχουν αντικειμενικά προβλήματα, τα οποία διαπιστώνονται, προβλήματα ρευστότητας, τότε να μπορούμε να δεχτούμε κάποιες ε, εξαιρέσεις για συμφωνίες business to business, αυτό ναι, αλλά σίγουρα η ευθύνη υπάρχει. Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται γρήγορα. Και συμφωνώ με την παρατήρηση που ακούσαμε για τους τόξους. Εγώ θα ήθελα να ξέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς βλέπει την ε, διαφορά των 40, των 70 ευρώ. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει περισσότερα πράγματα και ενδεχομένω να εξετάσει την περίπτωση αλλαγής. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Ιταλική ε, Γερουσία, στον κύριο Αντώνιο Παναβία. Το μικρόφωνο του είναι κλειστό, δυστυχώς δεν τον ακούμε. Σκούζα. Ζητώ συγγνώμη, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε για να σας μεταβιβάσω κάποιες σκέψεις ε, κάθε χώρας, την προβληματική κάθε χώρας και να θέσω στην προσοχή σας αυτά τα θέματα για τις αποφάσεις που θα λάβετε. Θέλω να κάνω διάκριση μεταξύ καθυστερήσεως πληρωμών και τρόπων πληρωμών. Στη χώρα μας, στην Ιταλία, αλλά νομίζω και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, από παλιά υπήρχαν διάφορες, διάφοροι τρόποι εξόφλησης και διάρκεια μεγάλη χρονική στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Εν γέννη κυμαίνεται μεταξύ 60 και φτάνει μέχρι 180 μέρες. Αυτή είναι ένας τρόπος πληρωμός, διάρκεια. Διαφορετικό πράγμα η καθυστερημένη πληρωμή. Λοιπόν, τα μέτρα που θέλετε να λάβετε, πρόκειται να λάβετε, σε σχέση με τις κυρώσεις που θα πρέπει να δημιουργηθούν για να γίνονται σεβαστές οι προθεσμίες πληρωμών είναι ένα θέμα. Μία βα... βαθμιαία εφαρμογή των μέτρων που θα θεσπιστούν χρειάζεται διότι σε κάποιες χώρες ίσως να έχουν κάποια αρνητική συνέπεια. Εγώ φαντάζομαι στις ταλικές επιχειρήσεις που έχουν διάφορες συμβάσεις και πολιετή συμβάσεις που προβλέπουν ε, προθεσμία πληρωμής μακρύ, μεγάλο, ενώ αντίθετα για τους προμηθευτές τους ισχύουν οι ίδιοι χρόνοι που ξαφνικά θα μπορούσαν να μειωθούν τα διαστήματα αυτά και να μειωθούν στις 60 ή ακόμα στις 30 μέρες οι προθεσμίες πληρωμής. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Σας θέτω λοιπόν την ανάγκη προβληματισμού επ' αυτού. Να γίνουν κατανοητοί τι λόγια λόγοι τους οποίους σε αυτές τις χώρες υπάρχουν μεγάλες προθεσμίες πληρωμής, ίσως και επειδή καθυστερούν να πληρώσουν και οι δημόσιες δικής σε αυτές τις χώρες. Να προσέξετε, θα πρέπει σταδιακά να εισαχθούν αυτά τα μέτρα που θα θεσπίσετε για να εξασφαλιστεί αυτή η ομοιομορφία που θέλουμε όλοι μας και εγώ εκπροσωπώ και τους Ιταλούς επιχειρηματίες. Και θα ήθελα μια συζήτηση με τις άλλες ε, σε σχέση μάλλον με τις άλλες χώρε, θα θέλαμε οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την εφαρμογή των νόμων είναι παρόμοιε. Υπάρχει ομοιομορφία. Ευχαριστώ. Θα δω το λόγο στην Πρόεδρο Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων ε, της, ε, του Λιθουανικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Ντένις Μπούντρι. Είναι εκεί. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πρόταση για οδηγία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές θα συμβάλλει στη διασφάλιση της λειτουργίας ε, ενός πολύ σημαντικού τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το έγγραφο αυτό αποτελεί μέρος της ατζέντα της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και αποτελεί μέρος ε, της πρωτοβουλίας Small Business Act, καθώς και του Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης της Ευρώπης. Όσον αφορά την συγκεκριμένη διατύπωση της συγκεκριμένης πρότασης, ε, θα ήθελα να εκφράσω τις θέσεις του Λιθουανικού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη ε, διατύπωση του άρθρου 4.1. Η Λιθουανία πιστεύει ότι ε, είναι σωστό να εγκρίνουμε την πρόταση με την εξή διαφοροποίηση όσον αφορά τα ποσά. Για χρέος ε, λιγότερο των 1.000 ε, ευρώ θα πρέπει η αποζημίωση να είναι 40 ευρώ. Για πάνω, άνω των 1.000 ε, ευρώ, 70 ευρώ να είναι το κόστος ίσπραξης και για ποσά 10.000 με 100.000 ευρώ το η αποζημίωση για την ίσπραξη θα πρέπει να ανέρχεται σε 200 ευρώ. Και όσον αφορά το άρθρο 5.5 ε, προτείνουμε 2% αντί για 5% ε, αποζημίωση. Επίσης, θα θέλαμε να συμφωνήσουμε με την 12η προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής ε, για την Οστερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών, ε, τον κύριο Μάρκον Χάρτο και την κυρία Μπάρβαρα Βάιλερ, για την διοργάνωση της σημερινής ε, συζήτησης που στόχο έχει τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Τελευταίος σκιώδης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κ. Ματέο Σαβίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω σε αυτά που είπαν αρκετοί προλαλήσαντες. Καταλαβαίνω αυτούς που έχουν δισταγμούς που λένε ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ. Μιλάμε και για θέσεις που χάνονται. Περίπου 450.000 θέσεις απασχόλησης υπολόγισε η ΟΚΕ ότι χάνονται λόγω καθυστερήσεως πληρωμών. Για μερικούς είναι οικονομική διαδικασία και συμβατική που ακολουθείτε. Οπότε είναι αμετακίνητη όσον αφορά τη Λέγα του Μπορά, η θέση της Λέγα του Βορρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σ' όσα λέει η οδηγία. Πέρα από το δημόσιο τομέα, που πρέπει να σέβεται το χρόνο πληρωμής, όπως συμβαίνει σε κάποιες χώρες όπως η Φιλανδία ή η Σουηδία, αυτομάτως θα πρέπει να επιβάλλονται τη για τις καθυστερήσεις, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη από πλευρά των μικρομεσών επιχειρήσεων, που δεν το σκέφτονται καν να το κάνουν, οι μεγάλοι διανομή χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα τη σύμβαση για να στραγγαλίσουν, αν θέλετε, τους προμηθευτές και να τους αποσπάσουν ε, τις καθυστερημένε πληρωμέ. Λοιπόν, και ο μεγάλος ιδιωτικό τομέα ε, ίσω ασκεί ένα ε, μονοπόλιο που δεν υπάρχει ούτε στο δημόσιο. Στην Ιταλία δεν είναι αποτελεσματικός ο δημόσιος τομέας. Και από την πλευρά ο ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ε, καμιά φορά ακολουθεί μονοπολιστική προσέγγιση, είναι ακόμα λιγότερο ακριβής στις ε, πληρωμές του. Και τώρα ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και Μηχανικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου της Αυστρίας, ο κύριο Κόνραντ Στάνταλ. Συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά το όνομά σα, δεν μιλάω γερμανικά. Κυρίε και κύριοι, η Αυστρία επικροτεί την πρωτοβουλία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε οικονομικά δύσκολου καιρού να υποστηρίξει ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα και τις απαραίτητες πιστώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χαιρόμαστε λοιπόν που προτείνονται εδώ συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων πληρωμών. Διαπιστώσαμε ότι ειδικά όσον αφορά τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ε, συναντάμε δυσκολίες που συνδέονται με τις καθυστερήσεις πληρωμών. Ιδιαίτερα ε, στις επιχειρήσεις εξαγωγής ξύλου που αποτελούν ε, σημαντικό τομέα στην Αυστρία. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν ευρωπαϊκά πρότυπα για τον τομέα αυτόν. Επίσης, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικό να βρεθούν πρότυπα συμβάσεων με τους παραγωγούς, ώστε και στο μέλλον να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που φαίνεται ότι θα επιδεινωθεί. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συναντούν σημαντικά προβλήματα χρηματοδότησης και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εγγύρες πληρωμές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, λοιπόν, για τα εθνικά κοινοβούλια, για το ευρωπαϊκό, δεν έχουμε άλλους που ζητούν το λόγο, τέσσερις γυναίκες έχουμε το Ευρωκοινοβούλιο. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ η κυρία Ροήτοβα, η κυρία Κόμι και η κυρία Γκέπχαρτ. Δύο λεπτά η κάθε μία. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, δεν ζήτησα το λόγο. Καλώς. Κυρία Ροΐτοβα, ζητήσατε το λόγο εσείς. Ναι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ όλο το δίλεπτό μου. Και εγώ πιστεύω ότι οι καθυστερημένες πληρωμές στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά και χρειάζονται αυτηρότερες κυρώσεις. Όχι μόνο επιστροφή του κόστους, αν επιβληθούν κυρώσεις. Η απλούστευση του κειμένου θα βοηθούσε και απλούστευση του συστήματος. Γιατί όσο έχει το κείμενο μου δημιουργεί προβλήματα. Δεν συμφωνώ με διαφορετικά, διαφορετικές κυρώσεις για επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα ε, και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, παρόλο που καταλαβαίνω ποιες σκέψεις οδήγησαν σε αυτό. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Νοσοκομείο. Το οποίο νοσοκομείο μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως καθαρισμού, μπουγάδας και μπορεί να, να... του δώσουν χίλια ευρώ αν καθυστερήσει η παράδοση. Αλλά αν καθυστερήσει ε, το νοσοκομείο σε μια πληρωμή πρέπει να πληρώσει πέντε φορές παραπάνω χρήματα. Δεν είναι λογικό αυτό. Θέλουμε να συνεχίσει η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Το νοσοκομείο είναι μια δημόσια υπηρεσία. Υπάρχει διάκριση λοιπόν μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και δεν είναι καλό αυτό και το 5% είναι πολύ ψηλό ποσοστό. Επίσης δεν συμφωνώ με το ότι το 5% δεν καταργείται μετά κάποιο χρονικό διάστημα. Ίσως μπορούμε να το αλλάξουμε και να το κάνουμε αργότερα 7% ή 10%. Από την πλευρά του καταναλωτή τώρα, αν κάποιος καθυστερήσει μια πληρωμή, Αυτός ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να αποζημιωθεί για κάτι που δεν πήγε σωστά την πρώτη φορά. Άρα νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας όσον αφορά αυτή την οδηγία. Ευχαριστώ. Κυρία Κόμη, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εισηγητές διότι είναι ένα θέμα ιδιαίτερα περίπλοκο και εδώ βλέπουμε και τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ κρατών μελών, που σίγουρα είναι σημαντικέ οι διαφορέ. Η ανησυχία μου ποια είναι ότι η οικονομική και η κρίση πολλέ φορέ περιορίζει τη δυνατότητα επενδύσεων και ταυτόχρονα αυξάνει όμω τα χρέη μέσω μακροπρόθεσμα. Οπότε οι πιο επιχειρήσει που πλήττονται περισσότερα και το βλέπουμε καθημερινά είναι εκείνε που είναι μικρέ και μεσαίε σε διάσταση, που όμω έχουν τη μικρότερη δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν δανειοληπτικέ δυνατότητε. Το να εισάγουμε μεγαλύτερη αυστηρότητα στον πληρωμών θα βοηθήσει τι επιχειρήσει να έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα και να μπορούν και στο μέλλον να κάνουν επενδύσει πιο σίγουρε τη στιγμή που θα έχουν την ασφάλεια ότι μπορούν να έχουν επιστροφή των χρημάτων τους. Ε, θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Πολύ συχνά, όπως συμβαίνει στην Ιταλία, το κράτος προσφέρει πρωτογενείς υπηρεσίες και αγαθά που έχουν πολύ πιο υψηλό κόστος, δημιουργούν ε, ταθητικό στον προπολογισμό μεγάλο. Ο ιδιωτικό τομέας έχει μεγαλύτερη ευελιξία. Ε, μάλλον λιγότερη γραφειοκρατία εν συγκρίση με το δημόσιο τομέα. Πιστεύω λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε χρονικό περιθώριο μεγαλύτερο στο δημόσιο τομέα και στον τομέα της υγείας συνεπώς. Τι ο τρόπος ίσως και η Ιταλία θα γίνει ε, πιο φρόνιμη χώρα διότι είδαμε ότι η χρόνια πληρωμή στην Ιταλία ε, είναι χρόνο που είναι η πιο προβληματική. Και ίσως αυτός είναι ένας τρόπος να βοηθήσουμε και τις χώρες που δεν είναι τόσο καλές και φρόνιμες όπως άλλες στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Γέπαρτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ε, τώρα θέλω να αναφέρω κάτι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για εμάς. Θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουν την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν. Εκ μέρους της ε, πολιτικής μου ομάδας ε, των Σοσιαλδημοκρατών ε, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι χρήσιμο στη συγκεκριμένη πρόταση να έχουμε διάκριση ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις μεγάλες διότι αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη σύγχυση και όχι σε καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Όσον αφορά το άρθρο 5.5 θα ήθελα εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας να πω ότι Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατυπωθεί με τρόπο πιο ε, σκόπιμο και πιο δίκαιο. Και ήθελα να το πω αυτό στην κυρία Βάιλερ. Ε, θα πρέπει να έχουμε μια διάκριση. Η καθυστέρηση μια ημέρα και ενό έτου ε, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Να δούμε πώ μπορούμε να βρούμε μια ρύθμιση πιο δίκαιη Ε, καλύτερο βέβαια είναι να μην υπάρχουν καθόλου καθυστερήσει πληρωμών, αλλά να βρούμε μια ρύθμιση σε περίπτωση που ο ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ε, καθυστερεί πληρωμέ του. Ο κύριο Κούλτσοτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι βουλευτέ, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Οι εμπορικέ επιχειρήσει πρέπει να ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώ είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν έγκαιρα τι οφείλε του προ το δημόσιο. Αλλιώς πρέπει να πληρώσουν πρόστιμα, αποζημιώσεις και βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Το δημόσιο προσφεύγει πολλές φορές σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θα έπρεπε και τότε το δημόσιο να πρέπει να πληρώνει έγκαιρα τα χρέη του. Καταλαβαίνετε ότι αλλιώ δεν μπορούν οι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει να πληρώνουν του ε, υπαλλήλου του όταν το δημόσιο καθυστερεί πάρα πολύ τι πληρωμέ του. 30 μέρε για μα είναι μια καλή περίοδο. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη προθεσμία αυτή μόνο στην περίπτωση που αμοιβαία έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο μεταξύ των δύο πλευρών και να μην είναι ποτέ πάνω από 60 μέρε. Το 60 να είναι το ανώτατο όριο για να γίνει πληρωμή. Το 5% τώρα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι από την πρώτη μέρα, αλλά να εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ισχύει και για μια μεγαλύτερη περίοδο. Τέλος, η πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις τροπολογίες των ε, βουλευτών πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να βοηθήσουμε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ σοβαρά προβλήματα με τις καθυστερήσεις πληρωμών. Όντως υπάρχουν χώρες που δεν αντιμετωπίζουν ε, ιδιαίτερα το πρόβλημα, αλλά άλλες πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και για να ολοκληρώσουμε το πρώτο τμήμα, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντς Πίτες Μάγερ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. κάποιους συλλογισμούς. Καταρχήν μιλάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εσωτερική αγορά. Τι, κανένα από τα δύο αυτά δεν είναι εναρμονισμένα στην εσωτερική αγορά. Εάν μια μικρομεσαία επιχείρηση ε, εκδίδει τιμολόγιο 50.000 ευρώ, δεν έχει σημασία αν ε, το τιμολόγιο αυτό ε, εκδίδεται για ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσια. Η μικρομεσαία επιχείρηση πρέπει να εισπράξει τα χρήματα αυτά. Δεύτερον, είναι πολύ, υπάρχουν πολύ διαφορετικές ρυθμίσεις ε, μέσα στην εσωτερική αγορά ε, σχετικά με τον ιδιωτικό τομέα και τον δημόσιο. Για παράδειγμα, έχουμε σε κάποιες χώρες ιδιωτικά νοσοκομεία, σε άλλες χώρες δημόσια ή και τα δύο. Ε, το νοσοκομείο είναι νοσοκομείο, ένα παράθυρο είναι παράθυρο, το τιμολόγιο είναι τιμολόγιο. Και όσον αφορά τους στόχους υπερημερίας, μιλάμε για αυτούς, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε η μικρομεσαία επιχείρηση τι τόκους πρέπει να πληρώσει στην τράπεζα για να γεμίσει το κενό από την καθυστέρηση μιας πληρωμής. Υπάρχουν ε, τα rankings, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ε, ε, ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά το, τους τόκους που πρέπει να πληρώνουν οι ίδιες. Ερώτηση λοιπόν, συλλογισμός, μήπως θα πρέπει η αντιμετώπιση μας ε, να σχετίζεται με το ύψος των τόκων και να μην έχουμε μια γενική ε, ρήτρα αποζημίωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το πρώτο τμήμα. Νομίζω ότι όσοι θέλησαν να πάρουν το λόγο τον πήραν. Τηρήθηκε ο χρόνος και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν και στο δεύτερο τμήμα και δεν ε, κάλυψαν όλο τους το χρόνο θα έχουν λίγο παραπάνω χρόνο. Τώρα ο Πρόεδρος της ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, Μπερναντέτ, που προείδρευσες με τόσο ωραίο τρόπο σε αυτό το τμήμα της συζήτηση, ε, Να συνοψίσω που βρισκόμαστε όσον αφορά τους ομιλητές, αλλά και όσον αφορά το λόγο που χωρίσαμε στα δύο τη συζήτηση, διότι όπως ξέρετε η μεγάλη κοινοτομία είναι αυτή που, ε, που βρίσκεται στο άρθρο 5. Εγώ και οι συνάδελφοί μου και κάναμε διάφορες συγκρίσεις και ξέρω ότι αρκετοί από εσά θέλετε να επανέλθετε να μιλήσετε ειδικά το θέμα αυτό. Έχω λοιπόν στον κατάλογο των ομιλητών κάποια μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που θέλουν να συζητήσουν για τα θέματα αυτά. Έχουμε χρόνο και για άλλους που θέλουν να παρέμβουν. Ε, τον κύριο Πρωτοπαπά σημειώνουμε, αλλά μπορείτε να μας ε, στείλετε και μία σελίδα. Ε, κύριε Κέπχαρτ, σας σημειώνουμε και τον κύριο Τρενταφυλλίδη. Παρακαλώ λοιπόν οι ευρωβουλευτέ ε, είτε να ζητούν το λόγο με τον συνηθισμένο τρόπο, οι συνάδελφοι από τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν ε, είτε να σηκώνουν τη ταμπέλα του είτε να μα ε, στέλνουν ένα χαρτί. Ο κύριο Ριπέιρο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε εκ μέρους του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου ε, θα ήθελα να ε, σας χαιρετήσω. Το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο συμφωνεί με τη σημασία της πρωτοβουλίας που συζητάμε. Για να έχουμε μια ισορροπημένη πρακτική ε, και έγκαιρη λύση δεν θα πρέπει να στηρίξουμε μόνο τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Δεν συμφωνούμε με τη διάκριση ανάμεσα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς διότι οι δημόσιοι φορείς πληρώνουν μεν αργά, αλλά στο κάτω, κάτω πάντα πληρώνουν. Ε, θα πρέπει να σκεφτούμε και την οικονομική συγκυρία που βρισκόμαστε. Ε, βρισκόμαστε τώρα μετά την κρίση, υπάρχει εμπιστοσύνη στο κράτος. Ε, εάν λοιπόν τώρα εισάγουμε διακρίσεις, στην πράξη θα συναντήσουμε σημαντικά προβλήματα για να για τη σταθεροποίηση του δημοσίου τομέα. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία το ποσοστό των 5% στις δημόσιες επιχειρήσεις επιχειρήσεις ε, θα σημάνει απώλειες ενός εκατομμυρίου μόνο για τον τομέα των φαρμακευτικών. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε οι διάφοροι φορείς να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους. Αυτό ισχύει και για, τους, ε, και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα. Για να μπορέσουμε να εισάγουμε τις αλλαγές αυτές ε, θα πρέπει να εισάγουμε ποινές όχι μόνο οικονομικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα για τις δημόσιες αρχές όπου είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις, ε, για παράδειγμα τόκοι υπερημερίας. Στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ειδών μέτρα μη οικονομικά. για την ε, πληρωμή χρεών από το δημόσιο. Στα τέλη του 2007 η προθεσμία πληρωμών από το δημόσιο μειώθηκε από 90 σε 60 μέρες. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, πρακτικές σας συμβουλές. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος αυτών των συζητήσεων. Ο κύριος Αχέρνα από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που οργανώσατε αυτό το φόρουμ για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Η αναδιατυπωμένη οδηγία για την καταπολέμηση των ε, καθυστερήσεων πληρωμών αποτελούν κεντρικό κομμάτι της ε, Small Business Act για την Ευρώπη ε, και για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επί της αρχής επικροτούμε κάθε μέτρο που θα βελτιώσει τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναγνωρίζουμε την σημασία διατήρησης των ροών πληρωμών και Συμφωνούμε με την ε, εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και την εισαγωγή ε, καλών, ε, καλής νοοτροπίας και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Η Ιρλανδία έχει εισάγει μέτρα για να διευκολύνει τις γρήγορες πληρωμές από πλευράς του δημοσίου. Το 2009 ο Αρμόδιος Υπουργός παρουσίασε μια πρωτοβουλία σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να ε, γίνεται ίσπραξη των χρηματων εντός 15 μέρου από την ε, παραλαβή του τιμολογίου. Τα αποτελέσματα όπως μετρήθηκαν το Δεκέμβριο ήταν πολύ θετικά. Το 91% των πληρωμών γίνεται εντός των 15 ε, ημερών και το 97% μέσα σε 30 μέρες. Τα νούμερα αυτά δείχνουν ε, πολύ υψηλό βαθμό συμμόρφωσης ε, για την εξασφάλιση των έγκαιρων πληρωμών. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν σημαντική πρόοδο και σημαίνουμε ότι το ότι αποζημίωση 5% είναι δυσανάλογη. Κλείνοντας, να σας ευχαριστήσω που οργανώσατε τη σημερινή συζήτηση που θα επιτρέψει η ανταλλαγή απόψεων για το σημαντικό αυτό θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αχέρν. Θα σας ενημερώσω σχετικά με τον κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Ευλίν Κέπχαρτ, κατόπιν η Πόλτη και η κυρία Κυρία Κέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ βρίσκω θετικό να έχουμε αυτή τη συζήτηση με, τα, με τους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, διότι είναι σημαντικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, ακούσουμε όλες τις διάφορες απόψεις, διότι η νομοθεσία μας ε, δεν ε, γίνεται αποκομμένη από, τους, από, τα γεγονότα στα κρατη Όσον αφορά τη διαφορά ανάμεσα στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ε, να πω ότι η πολιτική ομάδα ε, συναντά δυσκολίες στο θέμα. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει να γίνεται διάκριση του δημοσίου τομέα ε, στο θέμα αυτό. Είναι δύσκολο να το δει κανείς και κύριε Μάγερ έχετε δίκιο που είπατε ότι εντός της εσωτερικής αγοράς. Μιλάμε για εθνικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως ε, και συμπράξεις σε δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι φορείς αυτοί που ε, ανήκουν στο, σε όλο αυτό το σύστημα, στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Όσο περισσότερες διακρίσεις κάνουμε, τόσο πιο δύσκολο Ε, τόσο πιο ε, δυσνόητη γίνεται η νομοθεσία και γι' αυτό η πολιτική μου ομάδα είναι κατά της διάκρισης. Ευχαριστώ κυρία Κέπχαρτ, η κυρία Πόλτη, η κυρία Χίλε και ο κύριος Σβάμπ. Η κυρία Πόλτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι ξεκάθαρο ότι δεχθήκαμε πολύ θετικά την αναθεώρηση της οδηγίας για τη δυνατότητα, τη δυνατότητα επανεξέτασης της οδηγίας για τις καθημερινές πληρώμες. Στην Ιταλία διεξάγεται μια συζήτηση που υπογραμμίζει κάποια προβλήματα όσον αφορά την πρόταση οδηγίας και κάποιες απορίες όσον αφορά τους χρόνους που διατίθεται στη δημόσια διοίκηση δηλαδή 30 μέρες, θεωρούμε αντικειμενικά ότι είναι μικρό χρονικό διάστημα. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να έχουμε 60 μέρες ε, και να γίνεται πραγματικά σεβαστό αυτό το διάστημα. Διότι αντικειμενικά η δημόσια διοίκηση, οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να σεβαστούν αρχές διαφορετικές από αυτές από μια ιδιωτική επιχειρήση. Θα πρέπει ε, να με λειτουργικό τρόπο να κινηθούν ενώ ε, οι ιδιωτικές ε, δεν έχουν να λύσουν τα προβλήματα γραφειοκρατίας. Οι δικές μας περιοχές ε, και οι τοπικές διοικήσει έχουν να σεβαστούν το σύμφωνο σταθερότητα. Υπάρχει διπλή εντολή από την Ευρώπη. Πληρώστε γρήγορα τα χρέη σας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να προσέξετε να μην αυξήσετε τις δαπάνες γιατί παραβαίνετε το σύμφωνο σταθερότητα. Και αυτό για τη δημόσια διοίκησή μα είναι ένα πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά της καταποκοπήν κυρώσεις του 5% ε, αυτό μας δημιουργεί απορίες διότι φαίνεται σαν μια διάταξη που έχει ένα χαρακτήρα επιβολής κύρωσης, τιμωρίες και όχι ένα μέτρο που έχει χαρακτήρα, πώς να το πω, αποζημιωτικό όπως θα έπρεπε να είναι. Και αυτό όσον αφορά το δικό μας αστικό δίκαιο αλλά και όσον αφορά το αστικό δίκαιο που ισχύει και σε άλλες χώρες πιστεύω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Πέραν αυτού πιστεύω ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλα συστήματα για την επιβολή κυρώσεων κατά κάποιο τρόπο αλλά με μεγαλύτερη αναλογικότητα και μεγαλύτερη ευελιξία. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε. Σβάπ και Λορτ Μπάουνες μετά. Καλό, κύριε Σίκελεν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο τώρα στο δεύτερο γύρο. Και εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση να μην γίνει διάκριση ανάμεσα στις ε, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, και να ε, σας παρουσιάσω και ένα συλλογισμό. Η βασική αρχή της λειτουργίας ε, της εσωτερικής αγοράς είναι η ίση μεταχείριση. Εάν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε διάκριση χρειαζόμαστε πολύ καλά επιχειρήματα για να την ε, στηρίξουμε. Όπως άκουσα στη συζήτηση, κατά τη γνώμη μου δεν αρκούν τα επιχειρήματα για να στηρίξουμε την ε, τη διάκριση αυτή. Ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα. Όταν ακούμε όμως ότι το 90% ε, πληρώνει και μιλάμε μόνο για το 10%, δεν αρκεί αυτό για να τιμωρήσουμε τον δημόσιο τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό. Θα χρειαζόμασταν καλύτερα επιχειρήματα για κάτι τέτοιο. Και μην ξεχνάμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε και την καλή εικόνα του κράτους ε, ως ε, αναθέτουσας αρχής. Πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο να δώσουμε θετικά κίνητρα. Και ένα δεύτερο επιχείρημα γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εισπράξουν ε, τις οφειλές από, το, το, από τις αυτό όμως ε, δεν δικαιολογεί διάκριση σε σχέση με τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις, διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται ε, σε εξίσου δύσκολη θέση απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις, όσο και απέναντι στο, στις δημόσιες αρχές. Δεν αρκούν τα επιχειρήματα δηλαδή για διάκριση. Τέλος, όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις, ιδιαίτερα σε εποχές δημοσιοοικονομικής χρήσης, είναι δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να ε, λάβουν επιστώσει. Ε, γι' αυτό δεν δικαιολογείται η διάκριση ούτε στο τομέα αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χόγκλη, ο κύριος Σβάμπ και μετά ο Λόρδος Μπόουνες και ο κύριος Κουμπέρα, ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό οδήγησε σε πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε με την εισηγήτρια και τον σκιώδη εισηγητή μας Χάνσλικ. Ε, ε, ο νομοθέτης δεν έχει υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για να ε, θίξει το τις δημόσιες αρχές, αλλά για να αντικατοπτρίσει το γεγονός ότι ε, είναι κακοπληρωτή συχνά το δημόσιο και γι' αυτό δεν θα πρέπει να μιλάμε για διάκριση. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα οι Τελικά πάντως ε, είμαι της θέσης ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση. Δεν μιλάω για διάκριση δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε διακρίσεις, διότι έτσι θα έχουμε υπερβολικά ε, πολλές εξαιρέσεις μέσα στην εσωτερική αγορά. Το θέμα είναι τι κίνητρα μπορούμε να δώσουμε για να προωθήσουμε τις έγκαιρε πληρωμέ. και... Επίσης, όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, εάν δεν πετύχουμε τους, ε, Ο στόχος μας είναι να γίνονται έγκαιρα πληρωμέ. μήπως διευρύνουμε και στον ιδιωτικό τομέα τα σχετικά μέτρα. Αυτό το χρωστάμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δυστυχώς σε πολιτικό επίπεδο συχνά δεν ε, εκπροσωπούνται ε, επαρκώς θα δώσω το λόγο στον Λόρδο Μπόουνες, κατόπιν στον κύριο Κουμπέρα και τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Λόρδε Μπόουνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, φυσικά δεχόμαστε ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να πληρώνουν εγκαίρως λόγω των ε, χρηματικών ποσών για τα οποία μιλάμε. Αυτό μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην πρόθεση μιας κουλτούρας έγκαιρων πληρωμών. Εάν όμως πρόκειται να υπάρξει διάκριση θα θέλαμε να πούμε τα εξής. 30 μέρες προθεσμία μπορεί να μην είναι παράλογη δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει αυτό πρόβλημα για το δημόσιο τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Εθνικό Σύστημα υγεία, ε, που είναι ο μεγαλύτερο φορέας, πληρώνει το 90% των ε, τιμολογίων ε, μέσα στο διάστημα αυτό αλλά μέσα στον ενθουσιασμό μας να τιμωρήσουμε τον δημόσιο τομέα, να μην ξεχνάμε ότι οι ποινές, οι κυρώσεις αυτές ε, πληρώνονται τελικά από τους φορολογούμενους, όχι από κάποιον άσχετο φορέα ε, στον οποίο δεν ανήκουμε. Ε, είναι λοιπόν δυσανάλογη η ποινή του 5% ε, δεν έχει να κάνει με το... δεν λαμβάνει υπόψη πότε πληρώνεται τελικά η οφειλή. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, εάν είναι να υπάρξει ε, διάκριση, πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που λέει η συγγήτρια στο έγγραφο εργασία σχετικά με την πιθανή ε, συμπερίληψη των εταιριών ύδατος και ηλεκτρισμού. Δεν Ξέρω ποια είναι η διάκριση που γίνεται στην οδηγία που αναφέρεται στο σχέδιο αυτό του άρθρου, αλλά ζούμε σε έναν όλο και πιο ιδιωτικοποιημένο κόσμο, όπου πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν ε, τα καθήκοντα δημοσίων. Θα είναι λοιπόν ε, παράλογο να ε, αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής ε, που ισχύει για τις δημόσιες επιχειρήσεις ή ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτές που κάνουν τη δουλειά τους. Ευχαριστώ, Λόρδε Μπόνε, σε πολύ πρακτικές, σε πολύ ρεαλιστικές παρατηρήσεις. Ο κύριος Κουμπέρα, κατόπιν ο κύριος Τρινταφυλλίδη και τέλος ο κύριος Πρωτοπαπάς. Κύριε Κουμπέρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι εδώ ως γερουσιαστής Ταυτόχρονα από το 1994 και μετά ήμουνα δήμαρχος μιας πόλης 50.000 κατοίκων όπου πάντα ήταν ε, δεξιά η κυβέρνηση. Όχι μόνο πληρώνουμε έγκαιρα εκεί, αλλά δεν έχουμε ούτε πιστός ούτε χρέη. Και δεν θα τον ηρευόμασταν καν να παραγγείλουμε αγαθά υπηρεσίες και να μην πληρώσουμε έγκαιρα. Είναι κάτι φυσιολογικό για μας να πληρώνουμε έγκαιρα. Δεν χρειαζόμαστε οδηγία γι' αυτό. Αντίθετα, εμείς είμαστε πιστωτέ επιχειρήσεων που μας χρωστούν δεκάδες χιλιάδες τσεχικές κορώνες σε μισθώσει. Και αυτά τα χρέη δεν μπορούν να, να επιβάλλουμε την πληρωμή. Το άρθρο 5 γι' αυτό για μα είναι απαράδεκτο, διότι ε, ευνοεί ένα από τα μέρη. Ε, διερωτώ με πώς σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που καταπολεμά τη διαφθορά μπορεί να γίνει με τέτοια πρόταση. Πέραν αυτού μπορεί να είναι μια πηγή διαφθοράς όταν μιλάμε για συμβάσεις ενός εκατομμυρίου ευρώ. 5% σημαίνει 50.000 ευρώ, όπου μπορεί κάποιος υπάλληλο σκόπιμα να καθιστεί μια πυρομή, να δεχτεί μια ποινή, 3.000 ευρώ θα ήταν στη Τσεχία, τρεις φορές ένας μισθός και θα τσεπώσουν 10.000 ευρώ ε, σαν μερίδιο από ένα από τα συμβαλόμενα μέρη. Αυτό δεν είναι κακό. Άλλο αμφισβητήσιμο άρθρο είναι το άρθρο 10. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν κανένα εργαλείο να μπορέσουν να αποκτήσουν στοιχεία, λεπτομέρειες από, τις, ε, από τους ιδιωτικούς φορείς. Η οδήποτε λοιπόν έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας θα είναι ασφαλμένη και θα οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα. Αυτά συμβαίνουν, σημαίνουν ότι είναι ανεπαρκής ισχύουσα οδηγία. Και μόνο επειδή ανεπιτυχώς εφαρμόζεται δεν είναι ένας λόγος να τροποποιηθεί, κυρίως σε μια περίοδο κρίσεως όπου θα μπορούσε να είναι πιο επιβλαβής η οδηγία παρά εποφελής για κάποια κράτη-μέλη. Τεράστιες προσδοκίες μπορεί να σημαίνουν και μεγάλες τεράστιες απογοητεύσεις. Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση. Το βασικό πρόβλημα έγκυται αλλού. Κοιτάξτε τα κράτη-μέλη. Κοιτάξτε πώς πληρώνουν, πόσα χρωστάνε και πόσο άσχημα, πόσο πίσω έχουν μείνει όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Χάρμπουρ, ευχαριστώ για πολύ πρακτική άποψη που εκφράσατε κύριε Κουμπέρα. Ο κύριος Τριανταφυλλίδη και μετά ο κύριος Πρωτοπαπά, και μετά ο κύριος Σμούλεβιτς. Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε το λόγο. Όσο τρεις παρατηρήσεις. Εμείς σαν ομάδα της αριστεράς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πέραν από τις δημόσιες αρχές να στρέψει την πίεση της προς τις μεγάλες επιχειρήσεις με σημαντικά κέρδη. Αυτές κατέχουν μεγάλο μερίδιο στην αγορά και άρα διενεργούν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών έχοντας ταυτόχρονα και πολύ μεγάλο ποσοστό στις καθυστερήσεις των πληρωμών. Άρα στηρίζω και εγώ την άποψη για μεταφορά του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί βασικό χρηματοδότη των κρατών μελών. Η πολιτική πίεση προς τις δημόσιες αρχές για να συμμορφωθούν με τις καθυστερημένες τους πληρωμές θα πρέπει να συνοδευτεί με ανάλογα μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο ώστε και τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν έγκαιρα τη χρηματοδότηση που δικαιούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στην πίεση που δέχονται. Και τρίτο, στο εμπορικό κομμάτι, η εναρμόνιση των προθεσμιών πληρωμής για τον δημόσιο τομέα αφαιρεί ακόμα ένα διαπραγματευτικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αφενός δεν έχουν τους ανταγωνιστικότερους όρους κατά τη διεκδίκηση δημόσιων συμβάσεων, αλλά έχουν τη δυνατότητα ευελιξία στου όρου αποπληρωμή. Μια τέτοια ρύθμιση είναι σαφώ προ όφελο των μεγάλων σε μέγεθο επιχειρήσεων και θα οδηγήσει σε ενίσχυση τη μονοπωλιακή δύναμη του στην αγορά, αφού θα αποκλείσει από τι μικρομεσαίε τη δυνατότητα να προσφέρουν καλύτερου όρου κατά τη διεκδίκηση των δημόσιων συμβάσεων. Θα πρέπει λοιπόν, Πρόεδρε μου, να δούμε αυτό τον προβληματικό σημείο και να εξετάσουμε τρόπους αντιμετώπισή του. Ευχαριστώ. Uh, thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο κύριος Πρωτοπαπάς και μετά ο κύριος Μούλοβιτς και μετά ο κύριος Κρότσμαν. Παρακαλώ κύριε Πρωτοπαπά. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το θέμα των <coughs> δημοσίων υπηρεσιών, επαναλαμβάνω ότι η, τόσο η πρόβληψη για το δεσμευτικό όριο των 30 ημερών πληρωμής, όσο και η ποινή του 5% είναι εξαιρετικά αυστηρές έως υπερβολικά αυστηρές και νομίζω ότι σε αυτό το θέμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ε, επιπλέον, τίθεται ένα ζήτημα. Αναρωτιέμαι αν παραβιάζεται και η αρχή τη αναλογικότητα, διότι γίνεται διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και μάλιστα οφθαλμοφανής διάκριση και έντονη διάκριση, αλλά και επιβάλλεται ενιαία ποινή χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη διαφορά μεταξύ υγιών δημοσίων υπηρεσιών και αρχών που έχουν αντικειμενικά προβλήματα ρευστότητας. Θεωρώ ότι ε, το σχετικό άρθρο στι δημόσιε επιχειρήσει πρέπει να παρεξεταστεί στο σύνολό του. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνουμε τέτοια διάκριση και μάλιστα ιδιαίτερα αυστηρή διάκριση μεταξύ των ιδιωτών και του δημοσίου και να ε, λειτουργούμε δυσμενώ υπέρ του δημοσίου, εις βάρος του δημοσίου, ιδιαίτερα σε μια εποχή που όλοι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλές οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν προβλήματα, μεταξύ των οποίων και η δική μας και δεν το κρύβουμε, προσπαθούμε αντίθετα να τα θεραπεύσουμε και να βγάλουμε τη χώρα μας από αυτήν την κατάσταση. Αλλά βεβαίως ο δημόσιος τομέας εκ των πραγμάτων αποτελεί και ένα από τα κύρια εργαλεία για την ανάπτυξη και την τόνωση της αγοράς. Λοιπόν, ε, γι' αυτό το λόγο και διαφωνούμε με το σχετικό κομμάτι. Θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει και να αλλάξει ριζικά. Ε, θέλω τέλος να επισημάνω ότι ιδιαίτερα για τα νοσοκομεία και τους Δήμους στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα σε ασφιχτικές προθεσμίες και κάτω από τις φορούς συνθήκες. Uh, thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μούλοβιτς και μετά ο κύριος Κρότσμαν. Και μετά ο κύριος Πάσκο, που είναι και ο τελευταίος που έχω στον κατάλογό μου από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δεν ξέρω, υπάρχει κανένας άλλος από τα Εθνικά Κοινοβούλια που θέλει το λόγο. Α, κι εσείς, ναι, εντάξει. Ωραία λοιπόν. Παρακαλώ κύριε Σμουλίβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όσον αφορά το περιεχόμενο της πρότασης, πιστεύω ότι περιλαμβάνει πολλά σημαντικά πράγματα. Και στην αίθουσα αυτή ακούστηκαν επίσης πολλά σημαντικά. Εγώ θέλω να επιμείνω στα εξή δύο. Πρώτον, η προθεσμία των 30 ημερών για την πληρωμή. Στην περίπτωση σχέσεις μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του δημοσίου μου φαίνεται μια λογική προθεσμία. Διότι υπάρχει μια μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερη πρόσβαση, πιο εύκολη πρόσβαση χρηματοδότηση από πλευρά του δημοσίου τομέα. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να διευκρινιστεί περισσότερο είναι το θέμα των αποζημιώσεων όταν πρόκειται για το κόστος της ίσπραξης. Εδώ πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να ορίσετε καλύτερα το θέμα για να περιορίζεται η ελευθερία ερμηνείας του γιατί ποσό μιλάμε. Άπαξ και υπάρχουν ε, διαφορές, μπορεί να οδηγηθεί η υπόθεση στα δικαστήρια και τότε να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο η πληρωμή. Που σημαίνει ότι το σύστημά μας χάνει σε αποτελεσματικότητα. Επιμένω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για ποσά. Ο δημόσιος τομέας όταν καθυστερεί δύο-τρεις μέρες δεν θα έπρεπε να τυχαίνει ίδιας μεταχείρισης όπως συμβαίνει σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση για εβδομάδες και μήνες. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ο κύριος Κρότσμαν, ο κύριος Πάσκα και μετά ο κύριος Πονσιλίους που προσθέσαμε στον κατάλογό μας. Θα δούμε, μπορεί να μπορέσει κι άλλος ένας από τα Εθνικά Κοινοβούλια να πάρει το λόγο ενδεχομένως. Ο κύριος Κρότσμαν πάντως πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, στο γεγονός ότι η οδηγία αυτή στόχο έχει να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν διαβάσει κανεί την ερεύνα της Κομισιόν, βλέπουμε ότι ακριβώς αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα. Οι δημόσιες επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμό, λαμβάνουν πάντα χρήματα και στη Γερμανία συμβαίνει αυτό. εφόσον κινούνται εντό των πλαισίων του προπολογισμού τους. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά τις εξισώνουμε με τις δημόσιες, ε, τότε υπάρχει το πρόβλημα του πιστοτικού ορίου. Εάν το ξεπεράσουν, τιμωρούνται διπλά. Να αναφέρω τον κανονισμό Βασιλεία 2. Να τονίσω ότι Κανένας ε, δεν αναγκάζεται να απαιτήσει το 5% εάν ε, η καθυστέρηση πληρωμών ε, είναι μία ή δύο μέρες. Και επίσης να σας θυμίσω ότι σε όλη την Ευρώπη ισχύουν αυτά. Ο συνάδελφος από τη Ρουμανία μου λένε ότι στα νοσοκομεία πληρώνει μετά ένα χρόνο. Να μην αναφέρω καν την Ελλάδα. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα, αλλά ο στόχος μας είναι ακριβώς να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όσον αφορά την αποζημίωση. Φυσικά δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε ε, περιπτώσεις διαφθοράς, ε, όταν μιλάμε για το 5% ενός εκατομμυρίου. Ήδη όταν μιλάμε για 100.000, ε, το 5% είναι 5.000 ευρώ, είναι σημαντικό το ποσό, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μία οροφή ώστε και για το δημόσιο να μην είναι δυσβάστητα αυτά τα μέτρα αυτά. Το δημόσιο, αν πληρώνει, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να συμμορφωθεί με την οδηγία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κρότσμαν. Κύριος Πάσκα. Στο πήρα, στο πήρα. Πάσκα και μετά στο τέλο, η ε, κυρία Βερέν. Ο κύριο Πάσκα πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να σα χαιρετήσω και να χαιρετήσω και του άλλου εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι παρόντα και τα μέλη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, στο θέμα που συζητούμε. Αναφέρομαι τώρα στο άρθρο 5, πληρωμές που καταβάλλονται από τις δημόσιες αρχές. Η γνώμη της Επιτροπής μας στο, ε, στη γερουσία της Ρουμανίας είναι ότι η αρχή της συμβα... συμβασιακής ελευθερίας για την καταβολή των πληρωμών πρέπει να γίνεται σεβαστή. Σύμφωνα με τον νόμο στη Ρουμανία, το ποσό καταβάλλεται την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί από τα μέρη. Όταν δεν υπάρχει συμβατική υποχρέωση θα πρέπει να καταβάλλετε το τίμημα όταν παραδίδετε το αγαθό. Και στο άρθρο 1 της νομοθεσίας μας σχετικού νόμου στην Ρωμανία το επιτόκιο για τόκους υπερημερίες προβλέπει συγκεκριμένα. Και άρθρο 5 της οδηγίας λέει ότι τόκοι για καθυστερημένες πληρωμές μπορεί κάποιος να ζητήσει αποζημίωση κατά αποκοπή να ζητήσει 5% του οφειλωμένου ποσού. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι δυσανάλογο, έχει τη μορφή κύρωσης όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Συνεχίζω τις συζητήσεις για αυτό το άθρο. Πέραν αυτού, στη συζητήση στην Επιτροπή μας, έχουμε πρόταση Ρουμάνων βουλευτών που προτείνουν να εφαρμοστεί τροπολογία, τροποποίηση της οδηγίας. Δεν θα λάβουμε τελική απόφαση εμείς στο Κοινοβούλιο μας πριν λάβει τελική απόφαση το Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά την αναδιατύπωση της ε, παρούσης οδηγίας. Επόμενος, ο κ. Πόνσιλους, η κυρία Βερχέ και ο κύριος Ζωβέ Έχετε το λόγο κύριε Πονσιλούς. Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά σας. Σας ευχαριστώ, σωστά μας προφέρατε το όνομά μου. Νομίζω ότι η Πολωνία έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα προφέρουν το όνομά μου από ότι εσείς κύριε Πρόεδρε. Τέλος πάντων, Πρόεδρε, θα αναφερθώ εκ νέου στο άρθρο 2. Έχουμε σχετικά με αυτό την επιστροφή στο δημόσιο τομέα, την πληρωμή στο δημόσιο τομέα. Αν πρόκειται για τοπική αυτοδιοίκηση, για τοπική κυβέρνηση, ισχύει νόμος στην Πολωνία σχετικά με τους δημόσιους φορείς σε τοπικό επίπεδο. Αν κάποιος, παραδείγματο χάρη, οργανώσει δημόσια αγορά και δεν έχει χρήματα να καλύψει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τιμωρείται. Δυνάμει του ισχύοντος νόμου. Τώρα, νοσοκομεία, μουσεία, σχολεία και άλλα συναφή ιδρύματα Εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα. Στα νοσοκομεία η ρευστότητα είναι καμιά φορά πολύ προβληματική. Είναι ένα πρόβλημα πραγματικό που τίθεται εάν υπάρχει καθυστέρηση πληρωμής για υπηρεσίες που έχει παραγγείλει ο δημόσιος τομέας, ένας δημόσιος φορέας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Από τη στιγμή που ο δημόσιος φορέας δέχεται μία σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών και η πληρωμή καθυστερήσει, τότε προστίθεται ένας τόκος για την καθυστέρηση. Νομίζω ότι θα πρέπει όσον αφορά τους δημόσιους φορείς και τον ιδιωτικό τομέα να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Αυτή η οδηγία έχει στόχο την εξάλληψη της καθυστέρησης των πληρωμών. Ποιο είναι το πρόβλημα. Αν εισαγάγουμε τη λύση του 5% ανεξάρτητα αν η καθυστέρηση είναι μία μέρα ή πολλοί μήνες, αυτή η λύση δεν είναι λύση. Δεν επιλύει κανένα πρόβλημα. Κυρίως όχι το πρόβλημα που έχει σαν στόχο να λύσει η εν λόγω οδηγία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τη συμβολή των Εθνικών Κοινοβουλίων και κάποιοι συναδελφοί μου θα ήθελα να πάρω το λόγο, τους ενθαρρύνω να τηρήσουν το χρόνο τους, διότι χρειαζόμαστε και επίσης ε, και χρόνο για τη σύνοψη της ηγήτριας. Η κυρία Βερχέιν από την Περιφερειακή Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερως για το θέμα, ενδιαφέρεται για αυτή την πτυχή της δουλειά μας σχετικά με την οδηγία περί καθυστερήσεως πληρωμών, οπότε της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που έχω τη δυνατότητα να μιλήσω εκ μέρους της ε, Περιφερειακής Επιτροπής. Είναι σημαντικό να πάρουμε στα σοβαρά αυτά που ακούσαμε από αρκετές πλευρές. Ε, το θέμα της διάκρισης ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο και θα ήθελα εκ μέρους της Περιφερειακής Επιτροπής να ζητήσω ίση μεταχείριση πολλά προγράμματα που εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφερειών ε, σχετίζονται με τις δημόσιες προμήθειες ε, και η διαδικασία ανάθεσης είναι πολύπλοκη και σε... Ε, στην περίπτωση μεγάλων έργων είναι πολύ δύσκολο ε, να, να τηρηθεί η προθεσμία των 30 ε, ημερών. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία ώστε να μπορεί να παρατεθεί η προθεσμία στις 60 μέρες. Επίσης χρήσιμο θα ήταν να εξετάσουμε εκ των προτέρων εάν, είναι, ε, υπάρχει δυνατότητα στην οδηγία να εισάγουμε και τις πληρωμές με δόσεις Επικροτώ ότι ενισχύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσει με την οδηγία αυτή. Δεν νομίζω όμως ότι είναι χρήσιμο να γίνει διάκριση ανάμεσα στο δημόσιο τομέα ή στις μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Πολλές ε, προμήθειες γίνονται σε συνεργασία ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει η στις μεγαλες επιχειρησεις πολλε προμηθειε γινονται σε συνεργασια δημοσιου και ιδιωτικου Εμείς ως κοινοτικές αρχές ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα ε, για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Uh, much, Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τελευταίοι τέσσερις. Ζουβάν, Καράτσα Μπίλτ, Κόσιουσνικ και Ντιγιόνγκ. Αυτοί είναι τέσσερις τελευταίοι ομιλητέ στον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Τζουβάν τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθω σε μια παρατήρηση που έγινε από διάφορους συναδέρφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από τα Εθνικά Κοινοβούλια για το ζήτημα των εξαιρέσεων που ενδεχομένω θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές για ορισμένες υπηρεσίες που έχουν ε, έμεσους πόρους. Άκουσα για τα νοσοκομεία που συχνά η πληρωμή δεν γίνεται από τον ασθενή, αλλά από οργανισμούς ασφάλειες, κάτι το οποίο δημιουργεί ένα επιπλέον στάδιο στην ίσπραξη. Οπότε, οι οργανισμοί αυτοί δεν είναι δυνατόν με την ίδια ευκολία να υποβληθούν στους ίδιους κανόνες όπως και οι υπόλοιπε επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλουμε να έχουμε κατακαιρματισμό στους κανόνες μας. Ευχαριστώ. Uh, you. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι βουλευτής και στην προηγούμενη ζωή μου όταν ήμουνα στο Εθνικό Κοινοβούλιο δηλαδή, ε, από διάφορα μέρη, έζησα στην Ιταλία και ξέρω ότι όλοι ενδιαφέρονται για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις και θέλω να σας υπενθυμίσω σε όλους ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε μόνο για το δημόσιο τομέα και δεν είναι ο δημόσιος τομέας, είναι κυρίω οι μικρές και μισέ επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης και θα μας βοηθήσουν να βγούμε από την κρίση. Συμφωνώ και εγώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι το 5% είναι πολύ. Τώρα όταν μιλάμε για το δημόσιο, εδώ εξεπλάγει κάπως που άκουσα ορισμένους να μιλάνε για τιμωρία, για διακρίσεις κατά των φορολογούμενων. όχι, εδώ πέρα μιλάμε για έγκυρη πληρωμή στην ώρα της, τίποτα άλλο. Δεν βλέπω γιατί επειδή σε ορισμένες χώρες μας οι δημόσιες δικήσεις είναι άκαμπτες, καθυστερούν γι' αυτό και πρέπει και να το δεχτούμε. Όχι έχουμε μια ευθύνη απέναντι στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Δεν πρέπει να βάζουμε παραπάνω διοικητικό άχθος στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αντίθετα, αυτή η οδηγία θα πρέπει να βοηθήσει να δημιουργηθεί και μια νοτροπία έγκαιρης πληρωμής και να πιέσουμε για μέτρα κατά της γραφειοκρατίας, αντί απλώς να λέμε ότι θα την πληρώσουν οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Χωρίς αυτές δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τις καθυστερήσεις που οφείλονται στην κρατική γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Οι τελευταίοι δύο, Κόσιουσνες και Ντεγιόγκο τελευταίος. Κόσιουσνες πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω να κάνω κι εγώ μερικές παρατηρήσεις, παρακαλώ. Εδώ μιλάμε για μια οδηγία η οποία είναι ρυθμιστικής φύσεως και έχω μια ερώτηση. Είμαστε σίγουροι ότι αν κάνουμε τους κανόνες πιο αυστηρούς αυτό θα βοηθήσει. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος. Έπειτα, το θέμα της διάκρισης. Μιλάμε για τον δημόσιο τομέα, για τον ιδιωτικό τομέα και μιλάμε και για πληρωμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν οι δημόσιες αρχές αποφασίσουν να επενδύσουν στις υποδομές με τη βοήθεια των δημοτικών ταμείων, τότε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πληρώνει και πληρώνει μέσα σε 90 μέρες. Και αυτό δεν μου φαίνεται να τηρεί την αναλογία που θα έπρεπε. Αυτό λοιπόν που θέλω εδώ να υπογραμμίσω είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις. Το άρθρο 5 είναι ένα πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε να αποτελεί μέρος της οδηγίας. Ευχαριστούμε. Τέλος, ο κύριος Δεγιόνγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, με ρωτήσατε πριν αν ε, θα μπορούσα να μιλήσω για την Ολλανδία. Ναι, την έχουμε τη συζήτηση αυτή και στην Ολλανδία. Δεν μπόρεσαν να έρθουν οι συνάδελφοι, αλλά μα ενδιαφέρει πάρα πολύ στην Ολλανδία. Και όντω είναι κρίμα γιατί στην Ολλανδία έχουμε ένα σύστημα των 30 ημερών για την κυβέρνηση. Δεν έχουμε τα νοσοκομεία, δεν έχουμε τέτοιου είδου χρέη. Άκουσα του συναδέλφου που λένε ότι πρέπει να φροντίσουμε για τις μικρές επιχειρήσεις πάνω απ' όλα και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία την κρατική, να την περιορίσουμε στο ελάχιστα αναγκαίο. Έχουμε λοιπόν τις 30 μέρες όπως σας είπα, αλλά αυτό που θα έπρεπε εδώ να πούμε είναι ότι στο άρθρο 5 σημείο 4 αναφέρονται κάποιες εξαιρεσει οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να αποφύγουμε τις 30 ημέρες, οπότε αυτό είναι που θα έπρεπε να δούμε. Πρέπει να παραμείνει αυτό το σημείο εδώ ή όχι. Αυτός ο καθορισμός στο 5-4 πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι μόνο στην περίπτωση συμφωνίας business to business. Όταν δηλαδή μια μικρή επιχείρηση ενδεχομένω έχει κάποιες δυσκολίε, κάποια βεβαιότητα κτλ. κάποια συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου να μπορεί να το λύσει σε διμερή σχέση. Δεν θα πρέπει να είναι μια γενική εξαίρεση, αλλά θα πρέπει να προβλέπεται μόνο σε περίπτωση συμφωνίε business to business. Όσον αφορά τώρα το πρόστιμο του 5%, συμφωνώ ότι είναι αυθαίρετο. Ότι δεν υπάρχει διάκριση στο αν πρόκειται για καθυστέρηση μία ημέρα ή καθυστέρηση ενό μήνα. Οπότε θα έπρεπε και αυτό να το δούμε αναλογικά να πούμε 2% και μετά αν η καθυστέρηση παρατείνεται, τότε να αυξάνεται το ποσοστό. Ευχαριστώ. Well, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο, κυρίως τους επισκέπτες μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πολύ πλούσια ήταν η ανταλλαγή απόψεων. Κρατήσαμε πολλές σημειώσεις. Θα καλέσω σύντομα την κυρία Βάιλερ να συνοψίσει ακούγονται συνεισφορές της Επιτροπής Βιομηχανίας και της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Πριν από αυτό θεώρησα ότι θα ήταν καλό να ακούσουμε την κυρία Μπρίνκμαν που είναι η Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει την ευθύνη της προτάσεως που μας υπέβαλε και είναι τακτική επισκέπτη στην Επιτροπή μας. Ξέρω ότι δεν θα μπορέσει να καλύψει τα πάντα, αλλά είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε σε επαφή μαζί της άμεσα και το όνομά της μπορεί να είναι στα έγγραφα θα σας δώσουμε και το όνομα αν το έχετε. Κυρία Μπρίκμαν, το πολύ πέντε λεπτά για να αναφερθείτε σε κάποια από τα θέματα που θίγησαν στην πλούσια συζήτηση, ούτω ώστε να πάρουμε κάποια απάντηση από εσά και μετά θα προχωρήσουμε και θα ακούσουμε και τους εισηγητές και τους συντάκτες ε, γνωμοδοτήσεων. Έχετε το λόγο κυρία Μπρίκμαν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εν ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διοργάνωση αυτή τη συζητήσεω, πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα πολύ από τον πλούτο και το βάθος των αναλύσεων που παρουσιάστηκαν από κατά την άποψη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι συγκρατούμε εμεί από τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, μεγάλη, πολύ μεγάλη υποστήριξη όσον αφορά την πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει σαν στόχο πράγματι να δημιουργηθεί νέα νοοτροπία, νέο ε, πολιτισμό όσον αφορά την καταβολή των πληρωμών την έγκαιρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι ένα στόχο για σύγχρονη διοίκηση, οι επιχειρήσει και πιο συγκεκριμένα οι μικρέ και μεσέ επιχειρήσει να μπορέσουν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να ωφελούνται από την ενιαία αγορά υπό τις καλύτερες συνθήκες. Κάναμε κάποιες πολιτικές επιλογές που αμφισβητήθηκαν από κάποιους ομιλητές. Ένα από τα βασικά στοιχεία πιστεύω της συζητήσεως είναι η διαφοροποιημένη προσέγγιση. Γίνεται διαφοροποίηση όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων από τη μια μεριά και τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων από την άλλη. Πολλά ερωτηματικά εστιάστηκαν επ' αυτής της πτυχής. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις Εκφράσαμε στη μελέτη αντιχτύπου κάποιες από αυτές τις εξηγήσεις. Να επαναλάβω όμως εδώ ότι θεωρούμε ότι το βασικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια οδηγίας ενός μέσου ρυθμίσεως εναρμονίσεως ήταν αυτό το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που εξέφρασαν οι ίδιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ίδιες επιχειρήσεις. Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν το σοβαρότερο πρόβλημα είναι της καθυστερήσεως πληρωμών από το δημόσιο τομέα, τη δημόσια διοίκηση. Ήταν ομόφωνη αυτή η προσέγγιση και μας ζήτησαν να κάνουμε τα δέοντα μέσω νομοθεσίας. Και αυτό το στοιχείο της εναρμονίσεως της περίοδου πληρωμών είναι ένα στοιχείο εντελώς καινοτόμο εν συγκρίση με την ισχύουσα νομοθεσία, την ισχύουσα οδηγία. Βασιστήκαμε επί της εμπειρίας των κρατών μελών διαπιστώσαμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη οι 30 μέρες ήταν ο κανόνας ήδη, ακόμα και λιγότερο από 30 μέρες. Αντίθετα, ε, αλλού ξεπερνιέται αυτό το όριο. Θέλαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτή τη διαφοροποιημένη προσέγγιση και νομίζω ότι θα είναι σημαντικό στοιχείο για το μέλλον. Άλλες σημαντικότατες πτυχές που αναφέρθηκαν είναι το 5%. Είναι σαφές διαπιστώνω ότι υπάρχει ομοφωνία απόψεων πάνω σε αυτό, η οποία διατείνεται ότι δεν είναι ανάλογο μέτρο, δεν είναι αποτελεσματικό, ότι χρειάζεται μια προσέγγιση πιο ρεαλιστική. Ακούσαμε διάφορες λύσεις από την πλήρη κατάργηση, σταδιακή προσέγγιση, βαθμιαία προσέγγιση. Μπορούμε μαζί να προβληματιστούμε από αυτού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαθέσιμη να συνεργαστεί μαζί σας για την εξέβρεση μιας λύσης που θα, βρει, δίνει κίνητρα. Κίνητρα χωρίς το σύστημα να είναι υπερβολικό. Ζη, μας ζητήθηκε να εξετάσουμε και μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι ένα πρόβλημα αρκετά δυσεπίλητο στα πλαίσια εναρμονίσεως στα κράτη-μέλη και πρέπει να το προσέξουμε όλους ιδιαίτερος. Και πριν ξεκινήσουμε μια προσέγγιση που θα είναι τομιακή ή θα είναι ειδική, θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Ο ιδιαίτερος τομέας των δημοσίων νοσοκομείων είναι κάτι που εφήγει. Έχουμε επίγνωση ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στο συγκεκριμένο τομέα και είμαστε έτοιμοι και εκεί να προβληματιστούμε μαζί σας για να βρούμε μια προσέγγιση που θα λάβει υπόψη την εν λόγω ιδιαιτερότητα. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι 30 μέρες που προβλέπονται ως εναρμόνισης για την καταβολή πληρωμών από το δημόσιο τομέα, τη δημόσια διοίκηση, ότι προβλέπει και κάποιες παρεκκλήσεις, κάποιες εξαιρέσεις. Άκουσα πολλούς ομιλητές που μας ζητούσαν να είμαστε πιο σαφείς, να μην αφήσουμε ανοιχτή πόρτα στις παρεκκλήσεις και εδώ μπορούμε να συνεργαστούμε. Άκουσα επίσης έτοιμα για περισσότερη ευκαιρία για το πεδίο εφαρμογή. Και εκεί είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σα για να καθορίσουμε ξεκάθαρα το πεδίο εφαρμογή. Αυτά και σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ για την επικοδομητική σας ανταπόκριση. Θα συνεχιστεί η συζήτηση καθώς θα προχωρήσουμε στην διαδικασία εξέταση του θέματος στην Επιτροπή. Τι θα ήθελα να κάνω τώρα, να δώσω το λόγο στου δύο συντάκτε γνωμοδοτήσεω, στον κύριο Ντεάντζολη, καταρχά τη Επιτροπή Βιομηχανία, Ενέργεια και Έρευνα και στον κύριο Μπολισάρη, δύο λεπτά το πολύ ο καθένα για να αναφερθούν σε κάποια θέματα που του αφορούν και μετά θα δώσω το λόγο για να ολοκληρώσει και να συνοψίσει στην κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήδη δυνατόν και λιγότερο θα χρειαστώ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή, πρέπει να πω, ότι ήταν μια ωραία συζήτηση, διαφάνησαν διαφορετικές απόψεις και εξάλλου αυτό είναι φυσικό. 27 κράτη-μέλη, διαφορετικές καταστάσεις, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες. Ποια είναι η σύσταση. Εγώ δεν εισέρχομαι στην ουσία κάποιων ζητημάτων που χρειάζονται εμβάθυνση, ξεκινώντας από το πεδίο εφαρμογής, μετά να αντιμετωπιστεί το θέμα των σχέσεων δημόσιας διοίκησης με μικρές και μεσές επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις με μικρές και μεσές επιχειρήσεις και μετά το θέμα των κυρώσεων και το μέτρο του 5%. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία χρειάζονται ενδελεχή ανάλυση και να προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε και αυτά που υπόθηκαν στη συζήτηση μέσω μιας προτάσεως που πάνω απ' όλα θα είναι ισορροπημένη, αλλά θα έλεγα και αποτελεσματική. Εγώ θα έλεγα ότι όσον αφορά την εμβάθυνση για να βρούμε λύση, δεν θα πρέπει να λησμονούμε το στόχο που έχουμε για το, την όλη προσπάθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στόχος λοιπόν του νομοθετήματο είναι να προστατεύσουμε τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη καθυστερήσεω των πληρωμών. Διότι αν δεν δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, κινδυνεύουμε να κάνουμε να πεθάνουν πολλέ μικρέ και μέσα επιχειρήσει. Αυτό σημαίνει να πλήξουμε την οικονομία, να πλήξουμε την απασχόληση και την εργασία. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη το θέμα αυτό τη καθυστέρηση των πληρωμών και την ανάγκη ύπαρξη μια οδηγία που θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφή και πάνω απ' όλα αποτελεσματική και να προβλέπει και τα σωστά, να είναι έγκαιρη όσον αφορά την εφαρμογή τη και να προβλέπει σωστά χρονικά διαστήματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ αυτή, χρήσιμη αυτή η συζήτηση για να ακούσουμε τις διάφορες απόψεις και τις ευαισθησίες που διαφαίνονται από τις διάφορες χώρες μέλη. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο. Η οδηγία ε, γενικά αναγνωρίζεται σαν κάτι απόλυτα χρήσιμο, σαν κάτι αναγκαίο. Πιστεύω λοιπόν ότι η προβληματική των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι κοινή προβληματική για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ζητήθηκε και η προσοχή μας επί ενός σημείου. Αυτό ε, της της σχέσεως μεταξύ δημόσιας διοίκησης και ιδιωτικής, ε, ιδιωτικού τομέα. Να είναι ισότιμη η βάση. Στι σχέσει μεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων είμαστε στην δυνατότητα ελεύθερης, ελεύθερων συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, που είναι κάτι που αναγνωρίζεται στην Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να κινηθούμε εκεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πιστεύω όμως ότι όπως η αναφέρθηκε η δεσπόζουσα θέση κάποιων επιχειρήσεων έναντι άλλων, νομίζω ότι θα ήταν δυνατόν να φανταστούμε το να βάλουμε στις ρήτρε που είναι άκρως καταχρηστικές, τους όρους υπερβο... τις προθεσμίες πάρα πολύ μεγάλες που επιβάλλονται στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτικών εμπλεκομένων μερών και όχι μόνο στις σχέσεις μεταξύ δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα. Μπορούμε να εμβαθύνουμε σε αυτό για να γίνει πιο δίκαιη η σχέση μεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να σκεφτούμε ε, κατά πόσο είναι πολύ ισχυρό το ποσοστό που προτείνεται ακόμα και τη σχέση μεταξύ των ιδιωτικών τομέων όσον αφορά το 5% το μέτρο το αποτρεπτικό αυτό του 5% οι προτάσεις που ακούστηκαν από πολλές πλευρές μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο προσεκτική αξιολόγηση, ίσως και σε κάποια διόρθωση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Τέλεια. Τηρήσατε το χρόνο σας, πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας λέει ο Προεδρο. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Μπάρμπαρα Βάιλερ που νομίζω ότι έχει πολύ δύσκολη δουλειά. Ελπίζω να τα καταφέρει σε τέσσερα λεπτά να συναγάγει κάποια γενικά συμπεράσματα και ίσως ε, να δώσει κάποια ένδειξη για το μελλοντικό της χρονοδιάγραμμα, ούτω ώστε να ξέρουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Έχεις το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Μάκομ. Θα μπορούσα να το καταφέρω σε τέσσερα λεπτά, αλλά διαπίστωσα από τις παλές παρεμβάσεις ότι έχω ξεχάσει ένα σημείο και γι' αυτό θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για τη διάκριση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Καταρχήν όμως ε, να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ε, εθνικούς βουλευτές ε, και να σας επενέσω. Στην αρχή της σημερινής εκδήλωσης είχα την ανησυχία ότι θα παρουσιάσετε μόνο τις θέσεις των, Ευρωπαϊκών, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό δεν συνέβη και είναι σημαντικό αυτό. Τη θέση των ε, κυβερνήσεων σας ε, τις ε, λαμβάνουμε μέσω του Συμβουλίου και η σημερινή εκδήλωση είχε άλλο στόχο. Άκουσα λοιπόν μια σειρά πολύ ενδιαφέρουσων προτάσεων τις οποίες προλαβαίνω να συμπεριλάβω στην πρότασή μου όσον αφορά ε, το χρονοδιάγραμμα. Μπορώ να τις συζητήσω με τους κοιότητες συζητητές, πώς μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε, να τις λάβουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα. 27 κράτη-μέλη, 27 προτάσεις σχεδόν ακούσαμε. Θα πρέπει λοιπόν να ζυγίσουμε τι είναι εφικτό και τι είναι χρήσιμο. Ε, πιο εύκολο θα ήταν να υιοθετήσω την ε, θέση ε, του λιθουανικού ε, Δύσκολο θα μου ήταν να υιοθετήσω την ε, θέση της Λιθουανίας σε 2% αποζημίωση, αυτό μπορώ να το δεχτώ, αλλά την οροφή για την για την ε, αποζημίωση δεν μπορώ να τη δεχτώ, όπως επίσης ε, και τις προθεσμίες ε, για την εφαρμογή δεν τις βρίσκω πολύ ρεαλιστικές. Έχουμε μια οδηγία από το έτος 2000 η οποία δεν λειτουργεί όπως θα επιθυμούσαμε. Ε, εκεί ορίζεται ε, προθεσμία πληρωμών 30 ημερών χωρίς όμως καμία κύρωση και βλέπουμε ότι αυτό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Λίγο αποτέλεσμα τα είχε. Κάποια κράτη-μέλη έχουν εισάγει εθνικές διατάξεις οι οποίες λειτουργούν εξαιρετικά. Για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, οι κάτω χώρες, η Γερμανία μπορεί να αλλάξει η κατάσταση αν υπάρχει πολιτική βούληση. Υπάρχει ανάγκη για δράση, αυτό πιστεύω και χαίρομαι που συμμερίζεστε τη θέση μου. Ε, έχω αναφέρει κάποια θέματα, θα ήθελα όμως να σας αναφέρω τώρα γιατί πιστεύω ότι ε, ο δημόσιος τομέας ε, αποτελεί υπόδειγμα. Ακόμα και στην περίπτωση που στην ομοθεσία θεσπίσουμε την ίση μεταχείριση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ακόμα και αν το κάνουμε αυτό, που ακούσαμε ότι πολλοί το θέλουν αυτό, τότε παρακαλώ στη συζήτηση στις πατρίδες σας με τις επιχειρήσεις και με το δημόσιο τομέα να σκέφτεστε ότι ο δημόσιος τομέας έχει ε, άλλο ρόλο, έχει άλλες συνθήκες, ε, έχει προβλέψιμα και σταθερά έσοδα σε σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έχει η διαδικασία προϋπολογισμού, ε, σύμφωνα με την οποία μπορούν να ανατεθούν ε, ε, έργα εφόσον υπάρχουν στον προϋπολογισμό και όχι πιο πριν. Έχουν, έχει καλύτερη πρόσβαση σε πιστώσεις από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνήθως δεν έχουν προβλήματα ρευστότητας που έχουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Άλλο θέμα είναι οι δημόσιες προμήθειες όπου ορίζεται αρκετά αυστήρα πώς μπορούν να λειτουργήσουν οι μικρομεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Εάν ο δημόσιος τομέας πληρώνει εγκαίρος, όπως συμβαίνει σε αρκετά κράτη-μέλη, στη Γερμανία, στη Σκανδιναβία, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τον νόμο. Ήθελα λοιπόν να σας πω γιατί πιστεύω κάπως ότι υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες ε, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εισάγουμε τη διάκριση. Και επίσης ε, τώρα που θα επιστρέψετε στις πατρίδες σας, το 5% πράγματι απορρίπτεται, οι πληρωμές σε δόσεις παραμένουν ως έχουν. Θα φροντίσουμε να μην συμπεριληφθούν μόνο κυρώσεις στην νομοθεσία αλλά και θετικά κίνητρα. Δεν θέλουμε υπερβολικά πολλές εξαιρέσεις, δεν θέλουμε να μειώσουμε τα εθνικά πρότυπα και θέλουμε πρακτική νομοθεσία, θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργούν ε, θέσεις εργασίας, διότι αντιπροσωπεύουν τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να τις βοηθήσουμε να παραμείνουν καινοτόμε. Γενικά είναι πολύ πιο καινοτόμε από ό,τι πιστεύετε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι οι μεγάλε επιχειρήσει, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι που θα φέρουν την οικονομία μα εκεί που τη θέλουμε. Θα πρέπει λοιπόν να τι υποστηρίξουμε, να τι βοηθήσουμε και αυτό είναι το μήνυμα που λαμβάνω από τη, την, ε, από σημερινή εκδήλωση και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μπάρμπαρα πάρα πολύ. Έκανε πολλή δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα και ελπίζω όλοι οι συμμετέχοντες να θεωρούν ότι μπορείς να προωθήσεις αυτά που τόνισαν. Λοιπόν, Κάποιε σκέψει δικέ μου. Ο χρονισμό των συνεδριάσεων είναι κρίσιμη σημασία όσον αφορά τι επαφέ μα με τα εθνικά κοινοβούλια. Όπω είπε η Μπάρμπαρα Βάιλερ, είναι καθοδόν συντάξεω τροπολογιών. Είμαστε σε επαφέ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είδαμε την μελέτη αντιχτύπου, αλλά έχει τη σωστή χρονική στιγμή που διεξάγεται αυτή η συνάντηση για να τεθούν αυτά τα σημεία και έγινε και ακρόαση με τα μπλεκόμενα μέρη και τώρα είμαστε σε θέση να δούμε κατά πόσο η συγγήτρια μπορεί να καταλήξει σε ένα συμβιβασμό και κάποια πολιτικά συμπεράσματα. Ελπίζω βεβαίως ότι εσείς και οι κοινοβουλευτικές σας επιτροπές να συνεχίσουν τις επαφές μαζί μας, καθώς προοδεύει το θέμα, και ελπίζω να ενθαρρύνετε και τους συναδέλφους σας στις επιτροπές σας να κρατήσουν την επαφή μαζί μας. Ξέρω ότι προσεκλήθητε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποστείλετε προτάσεις για αυτή τη δουλειά και την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής Καλωσορίζουμε και αντίγραφα των προτάσεων που έχετε υποβάλει και έχουμε ετοιμάσει ένα ανθολόγιο αν θέλετε των προτάσεων. Δεν έχουμε παραλάβει όλε. Θέλουμε να, με τα χαρά να δεχτούμε τι δικέ προτάσει και να τι διαβιβάσουμε και στην εισηγήτρια. Θέλουμε και τα σχόλιά σα για αυτή τη συνεδρία, στη σημερινή, αν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μα. Πώ θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα. Θεωρούμε ότι είναι ένα απαραίτητο κομμάτι τη δουλειά μα αυτό. Έχουμε κάποια σχέδια σύντομα θέλουμε να διεξαχθεί άλλη μια τέτοια συνάντηση σαν ένα τμήμα ε, την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών ε, δεξιοτήτων. Θα σας στείλουμε ειδοποίηση πάνω σε αυτό και να σας πω, να σας υπενθυμίσω ότι όλη αυτή η συνεδρίαση ε, μετεδίδεται στο διαδίκτυο και θα δείτε στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου την ηχογράφηση, τη μαγνητοσκόπηση αυτής της συνεδριάσεως που έχετε στο σελίδες μπορείτε, θα χαιρόμασταν αν συμπεριλαμβάνατε στην ισοσελίδα σας την ομιλία σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αναφέρετε τη δουλειά που κάνουμε για να δείξουμε πώς συνεργαζόμαστε, διότι νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τους πολίτες. Να δουν οι πολίτες ότι και οι δύο πλευρές εργάζονται. Και αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε. Ευχαριστώ όλους ιδιαίτερω τους επισκέπτες μας που έκαναν ιδιαίτερη προσπάθεια να έρθουν εδώ να είναι μαζί μας για τις έξοχες συνεισφορές τους και ελπίζω να συνεργαστούμε εκ νέου στο μέλλον και ευχαριστώ ιδιαίτερος τους διερμηνείς για αυτό το πρώτο κτήμα της θα γίνει ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι λίγο πριν από τις 5.30 όπου θα ξαναρχίσει η τηλεδιάσκεψη με την ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Οι αδίποτε φίλοι μας θέλουν να μείνουν από τα Εθνικά Κοινοβούλια με τα χαράς να παραμείνουν στους παρατηρητές. Φοβούμαι ότι δεν θα σας επιτρέψουμε όμως να συμμετάσχετε. Ευχαριστώ ξανά που ήρθατε. Uh, ladies and gentlemen, we'd like to start the... Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε... Να ξεκινήσουμε τη διάσκεψη με την Γαλλική Εθνοσυνέλευση στις 5.30. Ε, βλέπω ότι βρισκόμαστε ήδη σε σύνδεση, βλέπω τους ε, συναδέφους μου. Ε, θα σας παρακαλούσα να εγκαταλείψετε ήσυχα την αίθουσα για να ξεκινήσουμε. Να παρακαλέσω όλους τους ε, συναδέρφους την ομάδα που θα συμμετάσχει να καθίσει. Διότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Και ναι, έχουμε κάποια ονόματα στον κατάλογο των ομιλητών. Θα σας παρακαλούσα τις ε, συζητήσεις σας να τις ε, διεξάγετε εκτός της αίθουσας, παρακαλώ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε σύνδεση. Μας ακούει το Παρίσι. I am receiving you actually. Ναι, σας ακούω. Να ξεκινήσουμε. Μάλκομ, να ξεκινήσουμε. Ρωτάει το Παρίσι. Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε, Πρόεδρε. Καλώς. Αγαπητέ Μάλκομ Χάρμπορ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα εκ μέρους της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων να χαιρετήσω τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Επιτροπής ε, ΙΜΚΟ, Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το 2010 πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ την Επιτροπή λοιπόν Εσωτερικής Αγοράς που δέχτηκε να οργανώσει αυτήν την ε, μεγάλη πρωτιά. Είναι πράγματι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια συνάντηση μεταξύ μας Εθνικού Κοινοβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με μια οδηγία η οποία συζητιέται αυτή την εποχή και αυτό μέσω βιντεοδιάσκεψης. Την πρωτοβουλία αυτή την αναλάβαμε για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε το διάλογο ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια μέσα στο νέο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας και Μάλιστα, όχι μόνο επειδή έχουμε την επικουρικότητα και την αναλογικότητα που μας αφορά μέσα, αλλά και ε, να συζητήσουμε και επί της ουσίας του κειμένου. Αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε ένα σημαντικό κείμενο για να εγκαινιάσουμε αυτή τη συνεργασία μεταξύ μας, μια που πρόκειται για πρόταση οδηγίας πολύ σημαντική για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Το κείμενο αυτό δημιουργεί βέβαια προσδοκίες, ελπίδες, αλλά και επικρίσεις. Θα συζητήσουμε λοιπόν πάνω σε αυτά Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας που ζητήσατε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη διάσκεψη. Μας γράψατε τον Οκτώβριο, χρειάστηκε κάποιο χρονικό διάστημα για να οργανωθούμε. Θεωρούμε όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση και σίγουρα η τεχνολογία θα λειτουργήσει άριστα σήμερα διότι τώρα έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει και η σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια έχει μεγάλη σημασία για μας. Από τη δική μας πλευρά είμαστε η πρώτη επιτροπή που το πραγματοποιεί αυτό. Ελπίζω ότι θα είναι μια ιστορική στιγμή όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Γαλλικής Εθνοσυνελεύσεως. Είναι πολύ κρίσιμη καμπή αυτή όσον αφορά την πρόταση. Θα ακούσετε αργότερα αυτά που θα πει η συγητής μας. Θα μιλήσει ο δικός της συγητής. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Σφαμπ, θα μιλήσει και οι σκιώδεις εισηγητές των πολιτικών ομάδων είναι στη διαδικασία προετοιμασία ε, προετοιμασίας μιας γνωμοδοτήσεώς μας και θέλουμε να ακούσουμε ποια είναι η δική σας άποψη από αυτού. Άρα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που μπορούμε να συζητήσουμε και να μιλήσουν ομιλητές και από τις δύο πλευρές και να ακολουθήσει η συζήτηση. Έχουμε μόνο μία ώρα. Ξέρω ότι η δική μας πλευρά έχει προγραμματίσει το χρόνο αγόρευση, είναι περιορισμένο, είμαι ότι έχετε κάνει το ίδιο, η κυρία Μαριέτα Καραμαλή, η συγγήτριά σα, θα ε, μας μιλήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, εισηγητές. Κυρίε και κύριοι, πριν μπω στο βάθο της συζήτηση στην ουσία, θέλω να συμπληρώσω κάτι όσον αφορά την οργάνωση τη συζήτηση αυτής. Είχαμε την ευκαιρία τηλεφωνικά να μιλήσουμε με τον κύριο Σφάκ, τον εισηγητή, και έτσι λοιπόν δεν θα θέλαμε ευθύ αμέσω να μπούμε στις λεπτομέρειες του κειμένου. Να εξετάσουμε δηλαδή τα διάφορα τεχνικά ζητήματα πρώτα απ' όλα το εύρος τους είναι τέτοιο και το περίπλοκο είναι τέτοιο που δεν νομίζω ότι θα μας έφτανε μία ώρα. Επίσης, συμφωνήσαμε εδώ στην ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση να ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση 2009, στη συνέχεια να, τον Νοέμβριο Επίσης παρουσιάσαμε μια ανακοίνωση και όλοι μαζί θα παρουσιάσουμε την άποψή μας σε μια τελική έκθεση. Όσον αφορά λοιπόν τα κύρια στοιχεία, τα απαραίτητα που θα αναφέρουμε, η ανακοίνωση της 5ης Μαΐου κατέληξε σε τρία στοιχεία απαραίτητα. Πρώτα απ' όλα εναρμόνιση στοχοθετημένη, δεύτερον ελαστικότητα υπερδοκρατών μελών ε, επειδή υπάρχει αρχή της επικουρικότητας και τρίτον ε, αυξημένη προστασία του καταναλωτή. Τα συμπεράσματα της έκθεσης του Νοεμβρίου επιβεβαίωσαν τα στοιχεία αυτά και τα ανέπτυξαν παρετέρω. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι ο στόχος είναι να διορθώσουμε δύο προβλήματα που υπάρχουν στο προτινόμενο κείμενο. Πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια, ακρίβεια, που οδηγεί σε αβεβαιότητες και κάποια ανασφάλεια νομικής φύσης αν θέλετε και έπειτα η ε, αυτόματη εφαρμογή θα οδηγούσε σε ένα επίπεδο όχι επαρκές προστασία του καταναλωτή. Μπορεί να φαίνεται παράδοξο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το κείμενο το οποίο προτείνεται ως ανώτατη προστασία. Τελικά προσθέτει στον καταναλωτή μια ελάχιστη προστασία, μια ελάχιστη ασφάλεια και κάλυψη. Πρέπει επίσης να επενθυμίσουμε εδώ ότι χρειάζεται και ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή που δεν αναφέρεται ως τέτοια στο κείμενο. Η ανώτατη δε προστασία απειλεί κάποιες διατάξεις που υπάρχουν στο εθνικό δίκαιο των χωρών μας. Και μάλιστα πιο συγκεκριμένα αναφέρεται κάποιο πρόοδος που έχει γίνει όπως η εξαποστάσεως ε, αγορά και πώληση και αναφέρονται και άλλα στοιχεία στη γραπτή έκθεση προς την ίδια κατεύθυνση. Επίσης μια ισοπαίδωση προς τα κάτω που εμείς δεν θέλουμε. Αυτό το σημείο ομόφωνα το συζητήσαμε και συμφωνήσαμε. Δεν πρέπει εδώ να επεκτιμάμε το ότι διακυβεύεται στο διασυνοριακό εμπόδιο, πρόκειται για ένα 7%. Οι εξαποστάσεις πωλήσει ε, επίσης και υπάρχει και το θέμα της γλώσσας και της απομάκρυνσης Όλα αυτά σημαίνουν ότι μπορεί να υπάρχουν διαμαρτυρίες, είτε τηλεφωνικές κτλ. Για να βελτιώσουμε λοιπόν το κείμενο και να καταλήξουμε σε ένα πραγματικό σημείο ισορροπία, πρέπει να κρατήσουμε μερικές βασικές αρχές και τι υπενθυμίζω. Ο στόχος μας να είναι υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Δεύτερον, να επικεντρωθεί το κείμενο στα βασικά σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και αναλογικότητας και έτσι να διατηρήσουμε τις αρμοδιότητες στα κρατημέλη εκεί που έχουν αρμοδιότητες και να προσαρμόσουμε στις προθεσμίες τα δικαιώματα του καταναλωτή και τις πρακτικές. Συνεπώς, να προβλέψουμε την εφαρμογή της αρχής της ε, ανώτατης προστασίας του καταναλωτή, εκεί όπου χρειάζεται και πρέπει, να είμαστε δηλαδή ρεαλιστές. Επίσης, να διευκρινίσουμε το εύρος εφαρμογής, το πεδίο εφαρμογής σε σχέση με άλλα κείμενα και το εθνικό δίκαιο και γι' αυτό έχουμε φτιάξει ένα πρώτο σχήμα. Πρώτα απ' όλα με κοινού ορισμούς διορθωμένους που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη αλλά που έχουν και τη δυνατότητα ενδεχομένω να επεκτείνουν την προβλεπόμενη προστασία και σε άλλες κατηγορίες πέρα των καταναλωτών. Οπότε θέλουμε δηλαδή να παραμείνουν ε, οι εγγύσεις που έχει παραπάνω η Έπειτα, κάποιες ε, γενικές πληροφορίες που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των συναλλαγών και στην εσωτερική αγορά και όσον αφορά τις ε, εξαποστάσεως συμφωνίες, ε, συμβάσεις που θέλουμε να ενισχύσουμε περισσότερο όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή. Επίσης, οι ειδικέ διατάξεις που έχουν να κάνουν με την εγγύηση αγαθών είναι κάτι αναγκαίο για να μην οπισθοχωρήσουμε να μην πάμε πιο πίσω, να μην είμαστε λιγότερο ελαστικοί. Όπως επίσης και για την ισχύ των μηχανισμών. Έπειτα για τις καταχρηστικές ρήτρες εμείς πιστεύουμε ότι ένας ευρωπαϊκός κατάλογος ενιαίος και τροποποιημένος από την Επιτροπολογία δεν είναι κάτι καλό. Προτιμάμε κοινέ ε, λίστες που όμως σταδιακά να εμπλουτίζονται από τους εθνικούς καταλόγους. Πριν σας δώσω το λόγο, ίσως θα έπρεπε ακόμα να δούμε κάποια θέματα όπως τι γίνεται με μελέτες αντικτύπου που ζητούν οι διάφορες ενώσεις καταναλωτών. Έπειτα μπορούμε να προβλέψουμε και κάτι όσον αφορά την εξέλιξη του δικαίου όσον αφορά την πραγματική ιδιοκτησία. Σας ευχαριστώ πολύ. Well, Ευχαριστώ πολύ για μια πλήρη εισαγωγή, κυρία Καραμαλή. Να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Αντρέα Σφάρπ, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να εκφράσω τη χαρά μου που βλέπω κάποιους συναδέλφους. Δεν μπορώ να τους δω, δω όλους, αλλά σύμφωνα με τον κατάλογο που έδωσε ο Προεδρο, υπάρχουν αρκετοί φίλοι τη εκλογική μου περιφέρεια από τα σύνορα μεταξύ Γαλλία και Γερμανία που είναι μαζί μα και είναι μεγάλη χαρά που σα βλέπω. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι Η κυρία Καραμανλή ανέφερε μια σειρά δισταγμούς ε, τους οποίους έχουμε λάβει υπόψη μας ε, στη δική μας Επιτροπή. Δεν είναι κάτι νέο, ούτε έχουν παρουσιαστεί μόνο από πλευρά ε, τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Έχουμε αποφασίσει την δουλειά μα πάνω στην οδηγία αυτή που έχω αναλάβει εγώ ω εισηγητή να η εργασία αυτή να γίνει ε, όσο γίνεται ε, σε συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η εσωτερική αγορά όμως ε, συνεχίζει να συναντά κάποια εμπόδια. Δεν θέλουμε καν να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια εσωτερική αγορά που να λειτουργεί τέλεια, αλλά το 7% του διασυνοριακού ε, εμπορίου που ανέφερε η κυρία ε, Καραμαλή μπορεί να αυξηθεί πιστεύουμε και γι' αυτό εξετάσαμε προσεκτικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξετάσαμε και τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου και διαπιστώσαμε ότι όχι μόνο η νομική αβεβαιότητα ε, στην αντιμετώπιση της οποίας θα συμβάλλει και αυτή η οδηγία, αλλά και οι γλώσσες και οι πληρωμές αποτελούν εμπόδια στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η πρόταση της ε, Επιτροπής πάντως προσπαθεί να εξαλείψει ένα εμπόδιο στο διασυνοριακό εμπόριο και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι σκόπιμη. Η εσωτερική αγορά και η προστασία του καταναλωτή, αγαπητοί συνάδελφοι, αποτελούν δύο όψεις του ιδίου νομίσματος ε, και γι' αυτό θα θέλαμε ε, εδώ στην Επιτροπή μας για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία του Καταναλωτή να επεξεργαστούμε με τέτοιο τρόπο την ε, πρόταση αυτή ώστε να πετύχουμε τις εξής προϋποθέσεις. Καταρχήν, βελτίωση της διασυνοριακής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών. Δεύτερον, υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή σε όλα τα κράτη-μέλη και τρίτον ε, να λαμβάνεται υπόψη η, η νομική τάξη των κρατών μελών ώστε να μπορούν ε, να επιλεγούν ευέλικτες λύσεις. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να ε, κλείσουμε κάποιους ε, τομείς, κάποια θέματα ε, και στο τέλος να γίνει μια μελέτη σκοπιμότητας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι σήμερα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να εξετάσουμε μαζί σας τα προβλήματα που βλέπετε από πλευράς του γαλλικού δικαίου. Η κυρία Καραμαλή ανέφερε κάποια από αυτά. Ε, θα θέλαμε δηλαδή να συζητήσουμε αυτά τα γαλλικά προβλήματα, τα προβλήματα της Γαλλίας. Φυσικά ως εισηγητής ε, κοιτώ την Γαλλία όχι μόνο μέσω βιντεοδιάσκεψης ε, και προσωπικά έχω σπουδάσει στη Γαλλία για παράδειγμα, έχω μείνει εκεί. από 27 κράτη-μέλη προέρχονται διάφορες παρατηρήσεις που, ακού, που ακούμε και ε, στόχος μας είναι να συνδυάσουμε τις παρατηρήσεις αυτές ώστε όχι μόνο οι κυβερνήσεις, μόνο οι επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές να μείνουν ε, ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο στόχος μου και γι' αυτό θα ακούσω με προσοχή αυτά που έχετε να πείτε ε, εσείς καθώς και οι συνάδελφοί μου της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σβάμπ. Ε, κύριε Λεκυγέ, ε, μας ακούτε καλά προτού να προχωρήσουμε στους σκιώδεις εισηγητές. 5 sur 5, pas de problème. Κανένα πρόβλημα, μια χαρά. Good. So, la technologie marche très bien aujourd'hui. Λοιπόν, η τεχνολογία πάει μια χαρά σήμερα. Καλώς. Θα συνεχίσουμε με παρεμβάσει των σκιωδών εισηγητών των διαφόρων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο καθένα θα έχει 1,5 λεπτό στη διάθεσή του για να παρέμβει και μετά θα ακούσουμε τη δική σα πλευρά και τη δική σα ομάδα. Η κυρία Γκέπχαρτ, που είναι η σκιώδη εισηγήτρια και συντονίστρια για την ομάδα S&D της Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκω κάποιους βουλευτές που γνωρίζω ήδη από τη δουλειά μου επί της οδηγίας υπηρεσιών και παλιούς ευρωβουλευτές από την πολιτική μου ομάδα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό να μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους. Θα μιλήσω γερμανικά τώρα, διότι θα μιλήσω για την οδηγία. Ε, ε, Αξιότιμοι συνάδελφοι, η πολιτική, μας η πολιτική μου ομάδα έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της οδηγίας αυτής και ε, έχουμε σημαντικά προβλήματα τα οποία αντικατοπτρίζονται και σε αυτά που είπε η κυρία Καραμανλή. Έχουμε πρόβλημα με την πλήρη εναρμόνιση που προβλέπεται. η οποία αφαιρεί από τα κράτη-μέλη κάποια δικαιώματα. Και τα δικαιώματα αυτά έχουν διαφορετική μορφή στα διάφορα κράτη-μέλη πλήρης εναρμόνιση είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στους πολίτες μας ε, και γι' αυτό η πολιτική μου ομάδα και αυτό αναφέρεται και στο ψήφισμα πατρί, ε, θέλουμε μία μεικτή προσέγγιση. Θέλουμε να δούμε πού υπάρχουν δυνατότητες εναρμόνισης, διότι αυτός είναι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ο καλύτερος τρόπος, αλλά και τα κράτη-μέλη να συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν δικό τους ε, δίκαιο το οποίο να προχωράει πιο πέρα. και ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, θα πρέπει να διατηρηθεί διότι αντιμετωπίζουν πολύ γρήγορα κάποια προβλήματα που προκύπτουν. Θέλουμε δηλαδή να αναπτυχθούν περαιτέρω τα δικαιώματα των καταναλωτών. Για να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να δεχτούμε πλήρη εναρμόνιση. Θέλουμε διατήρηση της ευελιξίας. Αυτή είναι η προσέγγιση μου. Ήδη ξεπέρασα το χρόνο μου, ζητώ συγγνώμη. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το θέμα, είναι δύσκολο να παραμείνει κανεί εντό του χρόνου ομιλία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέπχαρτ. Ο κύριο Ρομπέρο Φορ, που είναι ε, σκιώδη για την ομάδα Άλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι Γάλλοι στο Παρίσι αλλά και εδώ συνάδελφοι στι Βρυξέλλε και σε όλε τι χώρε τη Ενώση, είναι σίγουρο ότι αυτή η οδηγία δεν μπορεί να, μεταφραστεί σε επαναχώρηση από τα δικαιώματα των καταναλωτών σε όλα τα κράτη-μέλη της στη Γαλλία, στη Γερμανία και οπουδήποτε αλλού. Πιστεύουμε πραγματικά ότι το να δοθεί δυναμισμός στην εσωτερική αγορά ταιριάζει με αυξημένη εμπιστοσύνη που έχει ο καταναλωτής και για να έχει ο καταναλωτής υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης θα πρέπει να προστατεύεται σωστά και να μην αισθάνεται ότι αυτή η οδηγία θα είναι μια υπαναχώρηση όσον αφορά τα δικαιώματά του. Α είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν, θα πρέπει σήμερα να, θεωρήσουμε ότι, να θεωρούμε ότι οι συνοριακέ συναλλαγέ δεν είναι πολύ σημαντικέ, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται στο μέλλον. 5, 10 χρόνια, 20 χρόνια θα είναι πιο σημαντικέ συναλλαγέ αυτέ, κυρίω μέσω τη αναπτύξεως ε, του εμπορίου εξ και του διαδικτύου. Και γι' αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Η μέγιστη εναρμόνιση έχει σχετικά ένα πλεονέκτημα. Πιστεύω ότι την ημέρα που θα συμφωνήσουμε επί κάποιων κοινών πραγμάτων θα είναι δυνατόν να τα υλοποιούμε καλύτερα και να μπορούμε να ανταποκριθούμε στι προσδοκίε του καταναλωτού. Θα χρειαστεί και μία παιδεία για την κατανάλωση που θα διευκολύνει κάποια πράγματα με παρόμοια προσέγγιση να γίνουν τα πράγματα σε όλα κράτη-μέλη, υπό την προπόθεση ότι θα προηγούμεθα και θα συντονιστούμε με αυτά που έλεγα. Δηλαδή, να υπερασπιζόμαστε τον καταναλωτή και να μην υποχωρούν τα δικαιώματά του. Και χρειάζεται εναρμόνιση. Σε ποιο βαθμό, μέγιστη πιθανότατα σε πεδίο όπω είναι οι ορισμοί, το πρώτο κεφάλαιο, ίσω και στο κεφάλαιο 3, ακριβώ σχετικά με τι ε, πωλήσει και κατά τα λοιπά θα πρέπει ε, να είναι συμβατή συμβατοί οι ορισμοί σε κάθε χώρα της Ένωσης με το κοινοτικό πλαίσιο και γι' αυτό συμφωνώ με αυτή τη διατύπωση, δηλαδή της μέγιστης εναρμονίσεως, αλλά εξαιρετικά στοχευμένης εναρμονίσεως. Ε, Ευχαριστώ κύριε Ροσφόρ. Και τώρα για τους πρασίνους η κυρία είναι η συγγήτρια. Η Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο εκ μέρους ε, των Πρασίνων να πω ότι το σημείο κίνησης για μας ε, είναι ότι η οδηγία αυτή είναι οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Είναι λίγο μπανάλα, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει το επίκεντρο να είναι οι καταναλωτές. Μερικές φορές το ξεχνάμε στη διαδικασία αυτή νομίζω. Ως πράσινοι ε, δεχόμαστε το στόχο της πρότασης αυτής ε, να ε, ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά και να βελτιώσουμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία που να βελτιώσει την κατάσταση για τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Γι' αυτό θέλουμε να συμβάλλουμε επικοδομητικά. Έχουμε όμως και κάποιες επικρίσεις. Κάποια σημεία θα πρέπει να βελτιωθούν για να μπορέσουμε και εμείς να στηρίξουμε την πρόταση. Πιστεύουμε γενικά ότι είναι λάθος να εισάγουμε μηχανικά πλήρη εναρμόνιση στην οδηγία αυτή. Αυτό μάλλον είναι το βασικό μας παράπονο. Και γιατί τέσσερα πράγματα να αναφέρω. Καταρχήν, αυτό δημιουργεί ε, νομική αβεβαιότητα και ποιες είναι οι συνέπειες, ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής, ποιες είναι οι συνέπειες σε σχέση με το εθνικό δίκαιο. Άλλο θέμα, υπάρχουν ε, πολλά σημεία, όχι λίγα, όπου μειώνεται το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή σε όλη την Ευρώπη. Με αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τρίτον, αμφιβολούμε εάν θέλουμε να ενισχύσουμε το διασυνοριακό εμπόριο. Νομίζω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό προτού να ξεπουλήσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών για να προωθήσουμε τις πωλήσει. Να ε, εξετάσουμε δηλαδή τις συνέπειες Τη εφαρμογή τη οδηγία. Και τέλο, η οδηγία αυτή δεν ανταποκρίνεται στι απαιτήσει του μέλλοντος. Ε, κάποιοι αναφέρθηκαν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το μέλλον και αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην ε, οδηγία αυτή. Η οδηγία αυτή δηλαδή δεν κοιτάει το μέλλον. Θέλουμε αυτά τα τέσσερα σημεία να βελτιωθούν για να μπορέσουμε να στηρίξουμε κι εμεί την οδηγία. Uh, have... Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έντβαρ Κόζιστνικ που είναι σκιώδης εισηγητής της Ομάδας Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δράτω με τις ευκαιρίες και εγώ εκ μέρου της ομάδας μας να χαιρετήσω τους φίλους μας στο Παρίσι. Είναι πολύ καλή αυτή η δυνατότητα για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου τη κυρία Μπιέλαν, τη συναδέλφου που είναι η συγγήτρια ε, στην ομάδα μα. Μάλλον είναι σε μια εκδήλωση που σχετίζεται με το ολοκαύτωμα στην Πολωνία. Και εκ μέρους ομάδας μας να πω ότι οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί υποστηρίζουν πλήρη εναρμόνιση, πλήρη εναρμόνιση σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να περιορίσουμε τον κατακαιρματισμό του κανονισμού που ισχύει τώρα και θέλουμε να τονιστεί ιδιαίτερα η ενημέρωση των καταναλωτών. Και Συμφωνώ με τον συνάδελφο των Πρασίνων, το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αναφέρεται εκτενώς και νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να είναι κινητήρια δύναμη για την ίδια την εσωτερική αγορά. Αυτά και ευχαριστώ. Και για να κλείσει η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας την ΚΟΕ, ο κύριος Κυριάκος Τιανταφυλίδης. Κύριε αγαπητοί συνάδελφοι, ε, εκ μέρους της δικής μου ομάδας εγώ θα επικεντρωθώ στο βαθμό εναρμόνισης της προτινόμενης οδηγίας. Όπως έχει πει η συνάδελφος η κυρία Γκέιπαρτ των Σοσιαλιστών, η πλήρης εναρμόνιση που προτείνεται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ισοδυναμεί με ξεκάθαρη μείωση της προστασίας των καταναλωτών. Η πλήρης εναρμόνιση αφαιρεί από τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα που ανταποκρίνονται στις αντικειμενικές συνθήκες τη κάθε χώρα. Ιδιαίτερα στο τέταρτο κεφάλαιο που αφορά τις εγγυήσεις, η πλήρης εναρμόνιση μειώνει το εφιστάμενο πεδίο προστασία των καταναλωτών στις πλήστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει και από τη μελέτη που έχει διεξαγάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σύνολο των κρατών μελών. Ακόμα και στους τομείς που δημιουργεί νέο νομοθετικό πλαίσιο, αυτό αποτελεί πλέον την οροφή και η, διαδικα... και η δικαιοδοσία για τροποποίησή του μετατοπίζεται από τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, είναι ξεκάθαρο ότι με την εφαρμογή της πλήρους εναρμόνισης αυτοί που εποφελούνται τα μέγιστα από τη μείωση των διοικητικών κόστων είναι οι επιχειρήσεις. Εν τούτης δυστυχώς παρατηρούμε ότι η μείωση στα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων δεν συνδέεται σε κανένα σημείο της οδηγίας με μείωση του κόστους για τους καταναλωτές. Και κλείνοντα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια οδηγία στην οποία η προστασία των καταναλωτών περιορίζεται στο βαθμό που αυτή δεν επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και δεν προϋποθέτει επιπλέον κόστος για αυτές. Με αυτή την αρχή εμείς είμαστε αντίθετοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι η παροχή υψηλού επίπεδου προστασίας από τους εμπόρους προς τους καταναλωτές δεν αποτελεί μόνο δυνατότητα αλλά υποχρέωση για τις επιχειρήσεις. Uh, thank uh, um, Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ακούσατε διάφορες απόψεις των πολιτικών ομάδων, απόψεις των εισηγητών μας, οπότε θα σας δώσω τώρα το λόγο για να ακούσω τις απόψεις, να ακούσουμε τις απόψεις μάλλον των μελών της δικής σας επιτροπής. Καλώς θα δώσω το λόγο καταρχάς σε μέλη της σοσιαλιστικής ομάδας Ζερόμ Λαμπέρ και Ζαν Γκομπέρ Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρόταση οδηγία προβλέπει να αντικαταστήσει τέσσερι οδηγίε ελάχιστη εναρμόνιση, αυτή του 85 όσον αφορά τι πωλήσει εκτό επαγγελματική έδρα, αυτή του 1993 χωρί τι ρήτε καταχρηστικέ, του 1997 όσον αφορά τι πωλήσει εξ και του 1999 για τι εγγύσει αγαθών καταναλώσεω. Αντικαθιστώνται αυτέ οι τέσσερι μέσω μια οδηγία μέγιστη εναρμονίσεω. Όσον αφορά την ουσία η οδηγία του 2005 όσον αφορά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και τις μέγιστες εναρμονίσεως. Το ίδιο ίσχυε και με λιγότερες αποχρώσεις Προσπαθούσε η οδηγία του 2008 όσον αφορά τι πιστώσει προ του καταναλωτέ, όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντική αλλαγή που προσπαθούμε. Το κείμενο τη ελάχιστη εναρμόνιση του επιτρέπει να προβλέπουν εθνικά μέτρα πιο προστατευτικά για του καταναλωτέ. Αυτό έκαναν τα περισσότερα κράτη-μέλη. Αυτό το κείμενο επιτρέπει με ένα επίπεδο προστασία παρόμοιο να εκφράζει διάφορες ιδιαιτερότητες όσον αφορά τις ισχύουσες λύσεις. Δεν θα είναι πλέον αυτό εφικτό αν η μελλοντική οδηγία στο σύνολό τη έχει σαν στόχο τη μέγιστη εναρμόνιση. Ε, ήδη το, Απρίλιο του 2009 και Ιανουάριο του 2010 όσον αφορά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν αφήνουν αμφιβολίες. Λοιπόν, τα συμπεράσματά μας είναι κατά της μηχανικής εφαρμογής της αρχής της μέγιστης εναρμονίσεως σε έναν τομέα τόσο ευρύ όπως είναι αυτός που καλύπτεται από το κείμενο, διότι θα μείωνε κάτι τέτοιο το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Αυτή η αρχή της μέγιστης εναρμονίσεως θα επέφερε την κατάργηση κάποιων διατάξεων ρυθμιστικών εθνικών που εξασφαλίζουν μια προστασία ε, που ο καταναλωτή δεν θα ήθελε να παραιτηθεί από αυτή την προστασία. Θα ίσχυε αυτό για κάποιε προσυμβατικέ πληροφορίε, για την εγγύηση που παρέχεται στα αγαθά ή τι καταχαριστικέ ρήτρε. Άρα θα δημιουργούνται πολλά προβλήματα δεν θα πρέπει να μελούμε ότι το δικαίωμα της κατανάλωσης είναι το δικαίωμα και της εγκύτητας, το δίκαιο της εγκύτητας. Θα μπορεί να κανείς να, παρέμβει, να παρέμουν τα κράτη-μέλη για να τα αποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες που αντιπροσωπεύονται την προστασία του καταναλωτού και να ανταποκριθεί στις προσδοκίε τη κοινωνία. Τώρα εδώ όλα θα ρυθμίσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να ισχύει καλύτερα, να εφαρμόζεται καλύτερη αρχή τη επικουρικότητα και δεν θα πρέπει ε, να ε, να είναι τόσο εξελίξιμο ο νόμος. Δεν είναι ρεαλιστικός ο νόμος ε, στην πράξη. Ομοιόμορφος νόμος που θα υποθέτει ότι δεν υπάρχει καμία παρέκκληση όσον αφορά την ε, προστασία. Είμαστε σε ευαίσθητο τομέα και κάθε υπόθεση ε, παρέκκληση είναι κάτι που δεν μπορούν να αποδεχτούν οι κυβερνήσει και οι καταναλωτέ. Άρα είμαστε υπέρ μια προσεγγίσεω ρεαλιστική που θα βασίζεται σε μια εναρμόνιση μέγιστη, η οποία όμω θα είναι στοχευμένη πραγματικά, δηλαδή θα εφαρμοζόταν στα όσα είναι απολύτω αναγκαία. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο προσεγγίσεις μπορούμε να έχουμε όσον αφορά την κατανάλωση. Το ένα είναι εσωτερική αγορά και το άλλο είναι προστασία των καταναλωτών. Για μας δεν έρχονται σε αντίθεση το ένα με το άλλο, είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι το κείμενο δεν βασίζεται στην καλή ισορροπία ανάμεσα στι δύο αυτές προσεγγίσει και νομίζω ότι με αυτό συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όπω επίση και η Κομισιόν, αλλά και ενώσει των καταναλωτών που θεωρούν ότι το κείμενο ευνοεί τι επιχειρήσει. Τεχνικά μιλώντα, υπάρχουν δύο πράγματα που μα πήγαν πίσω. Το ένα είναι όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο. Το είπαν αυτό και οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μην επανέλθω. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το εθνικό δίκαιο και επίση το είπαμε εξαιτία αυτή τη αρχή τη μέγιστη εναρμόνισης. Πολλέ εθνικέ διατάξει απειλούνται. Κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό η επιχειρηματολογία που οδηγεί σε αυτές τις αποφάσεις δεν πείθει. Εγώ πιστεύω ότι δεν βοηθούν τα δικαιώματα του καταναλωτή σε περίπτωση διαμάχης. Πηγαίνουμε περισσότερο προς τα πίσω αντί να έχουμε πρόοδο. Η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δεν μπορεί να βασίζεται παρά μόνο σε έναν ελεύθερο ανταγωνισμό και θεμητό ανταγωνισμό, όχι αθέμητο. Άπαξ και δεν υπάρχει αρκετά καλή ποιότητα, αυτό πιστεύω ότι μας πάει πίσω ότι να μας πηγαίνει μπροστά. Ευχαριστώ. Merci. ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στα μέλη της ομάδας UNP, Λίζο Φουά, που αντικαθιστά τον Ντανιέλ Πασκάλ, που είχε πρόβλημα με το τρένο, Ζεράρ Βουαζά και Βαλερή Ροζό. Για δύο λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντική και οδηγεί σε ενδιαφέρουσες προόδους. Γι' αυτό είναι εξίσου σημαντικό να αναλύσουμε από κοινού τα σημεία που θεωρούμε που είναι ασαφή, κυρίως το πεδίο εφαρμογή είναι αυτό, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε λοιπόν το κείμενο, το ξεκαθαρίσουμε και θα πρέπει να κάνουμε δουλειά όσον αφορά τους ορισμούς Και για να μην μπούμε σε τόσε λεπτομέρειε τώρα σε αυτή τη φάση, θα ήταν ενδιαφέρον και σημαντικό να ακούσουμε ποιε είναι οι σκέψει σα επ' αυτού. Δεν μπορούμε έτσι αφηρημένα να ακολουθήσουμε κάποια λογική σε αυτή τη φάση. Θέλαμε να ακούσουμε κάποιε παρεμβάσει ήδη όσον αφορά να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στα 27 κράτη-μέλη. Θα μπορούσατε σε αυτή τη φάση να μα ενημερώσετε ποια είναι τα ερωτηματικά σα όσον αφορά τις υπηρεσίες διότι ορίζονται αρκετά ευρέω στη συνθήκη, στις διατάξεις για την ελεύθερη παροχή, όπως και στην οδηγία περιπηρεσιών. Πιστεύετε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τον ορισμό των προϊόντων που αφορά τα αγαθά της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των αγαθά, ε, τα διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το άλλο πλαίσιο όσον αφορά τους διαγωνισμούς, τις δημοπρασίες μέσω διαδικτύου, εκεί συζητείτε το θέμα, διότι Έχουμε την πληροφορική που παρεμβαίνει. Η συνάδελφος Μαρία Τακαραμαλή στην έκθεσή της, στην ομιλία της παρενέβη λέγοντας ότι ε, πρέπει να έχει δικαίωμα ο καταναλωτής μέσω του διαδικτύου να έρχεται σε επαφή με έναν επαγγελματία αλλά να έχει τα ίδια δικαιώματα όπως και κάποιος που συναλλάσσεται με τον κλασικό τρόπο εκτός διαδικτύου. Και το δικαίωμα της υπαναχώρησης, το δικαίωμα ε, αυτό ε, όσον αφορά τις δημοπρασίες, κατά πόσο θα περνά η πιο καλή προσφορά. Έχετε κάποια άποψη να μας κοινοποιήσετε ούτως ώστε να μπορέσουμε να παρατείνουμε τις ανταλλαγές απόψεων πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα πεδίο εφαρμογή αρκετά ευρύ που έχει να κάνει με όλε τι συμβάσει που έχουν να κάνουν με την κατανάλωση, ε, με αντικείμενα, με υπηρεσίε. Αυτό βέβαια δημιουργεί δύο προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, δύσκολα αντιλαμβανόμαστε τη σχέση με άλλες κοινοτικέ οδηγίες που εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση και υπάρχουν και πολλές. Δεν πρόκειται μόνο για το μεκά κείμενο όπως είναι για τον ή για τις οικονομικές υπηρεσίες, αλλά πρόκειται και για εγκάρσια κείμενα όπως είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες και κυρίως η οδηγία για τις ορισμένες πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου που έχουν να κάνουν με συμβάσεις οι οποίες μέσω διαδικτύου συνάπτονται. Έπειτα υπάρχουν και άλλοι τομεί που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένε δυσκολίε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γνωρίζει, μια που προτείνει διατάξει με πολλέ εξαιρέσει και χωρί να είναι σαφέ το πεδίο εφαρμογή. Έτσι έχουμε ένα κείμενο που δεν είναι πλήρε. Στο στάδιο αυτό δεν έχουμε κάποια βεβαιότητα για το ζήτημα αυτό θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε τις δικές σας απόψεις για ορισμένους τομείς που από ό,τι φαίνεται αποτελούν αντικείμενο ειδικότερη εξέτασης, ακριβώς επειδή ε, προβλέπονται για αυτούς κάποιες εξαιρέσεις. Εδώ έχουμε εντοπίσει τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα ακίνητα, την διοκτησία όσον αφορά δηλαδή την οικοδόμηση ή την ενοικίαση και για τα κτίρια γενικά έχουμε ένα ειδικό καθεστώς με δεκαετή εγγύηση. Έπειτα έχουμε και τις μεταφορές και εκεί υπάρχουν ειδικά κείμενα, ενώ πρόκειται για διαφορετικές πτυχές κάθε φορά. Ίσως εσείς από τα δικιά σας την πλευρά να έχετε εντοπίσει και άλλους τομείς πάνω στους οποίους θα έπρεπε να σκεφτούμε ειδικότερα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ανάμεσα στα θέματα που ακόμα δεν εξετάσαμε είναι ένα το οποίο αναφέρθηκε σε κοινοτικό επίπεδο κυρίως στα πλαίσια ομάδας εργασίας προπαρασκευής του Συμβουλίου και πάνω σε αυτό θα πρέπει να τοποθετηθείτε. Είναι των κοινωνικών υπηρεσιών. Είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πέρσι στα πλαίσια μέσα εκθέσεως που καταρτήσαμε τρεις συναδέλφους όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες, κοινοφελείς υπηρεσίες. Μπορέσα να προσμετρήσω ότι στην Ευρώπη όσον αφορά αυτό το θέμα ε, υπήρχε μεγάλη ποικιλομορφία και είναι ένα παράδοξο πέρα από αυτή την ποικιλομορφία να παρουσιάζουμε κοινωνική φυσιογνωμία που να μας διακρίνει από τον υπόλοιπο κόσμο και κυρίως εναντί τον ΗΠΑ. Ποιο είναι το συμπέρασμα που απορρέει και δημιουργείται στο πνεύμα. Ότι μόνο ο σεβασμός της αρχής επικουρικότητας επιτρέπει να σεβαστούμε αυτή την ποικιλομορφία και τις ιδιαιτερότητες καθενός από εμά. Όσον αφορά την ουσία, με μεγάλο προβληματισμό μαθαίνουμε ότι δεν εξυπακούεται ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες ήταν εκτός πεδίου εφαρμογή. Κατά την άποψή μα, οι κοινωνικέ υπηρεσίε παρέχουν υπηρεσίε που δεν απευθύνονται στον καταναλωτή, αλλά σε ένα ιδιαίτερο κοινό, εύθραυστο κοινό, για να καλύψει ειδικέ ανάγκε με κοινωνικού στόχου, κοινωνική συνοχή, ένταξη στην αγορά εργασία κλπ. Είναι κανόνε πιο ιδιαίτεροι από ότι εφόσον οι δικαιούχοι των υπηρεσιών δεν είναι πάντα σε επαφή με τον πάροχο πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά σε μια σχέση τριγωνική μέσω της παρεμβάσεω ενό τρίτου δημοσίου φορέα ε, τοπική αυτοδιοίκηση, είτε για το να καλυφθεί το κόστο, ή όπως την περίπτωση της παιδείας και της κατάρτισης για να πλαισιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Πιστεύω αυτό το στοιχείο θα πρέπει σαφώς να μην δημιουργεί αμφιβολίες, να είναι ξεκάθαρος και δεν θέλουμε εξαίρεση ή αποκλεισμό από το σώμα του κειμένου διατάξεις που θα δίνουν την εντύπωση ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο ότι ε, ε, θα μπορούσε να υπάρξει μια ένταξη συμπερίληψη μέσω πολιτικής επιλογής. Ευχαριστούμε για τα ειδικά θέματα που θέτει τώρα η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Θα δώσω το λόγο στον Γκόμες, στον τη Σεζούρ από το Νέο Κέντρο και βέβαια στην εισηγήτρια. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι διατάξει όσον αφορά τι ω αγορέ είναι οι πιο σημαντικέ όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Γιατί αυτέ θα επηρεάσουν τις διασυνοριακές συναλλαγές και η Επιτροπή μας λυπάται που πρόκειται μόνο για ένα 7%. Δεν μπορούμε φυσικά να εξαντλήσουμε το θέμα, δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, όμως θα επενθυμίσω ότι πιστεύουμε εμεί ότι πρέπει να διορθώσουμε σε αυτό το στάδιο. Επί της ουσίας πρώτα απ' όλα πιστεύουμε ότι χρειάζονται υποχρεώσεις για ειδική ενημέρωση όσον αφορά το τι προβλέπεται στο κείμενο. Δηλαδή να προβλέψουμε την υποχρέωση ε, ε, ε τηλεφώνου επικοινωνία, ώστε να μπορεί ο καταναλωτή να επικοινωνήσει. Για θέματα τώρα πολύ συγκεκριμένα, το γαλλικό δίκαιο που είναι και πρόσφατο, είναι ο ΑΤΕΛ του 2008, δεν φύγεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά το επίπεδο αναρμόνησης και κατά συνέπεια όσον αφορά την αρχή της μέγιστης αναρμόνησης. Πρέπει να αφήσουμε δηλαδή στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν νέες καταστάσεις προβλέποντας ρυθμίσεις που προσαρμόζονται σε αυτές τις νέες συνθήκες. Διότι οι καταναλωτές έχουν διαφορετική σχέση ανάλογα με την εγκύτητα που έχουν με την αγορά. Και αυτό έχει να κάνει και με τις προθεσμίες επίσης. Επί της ουσίας πάλι. Δεν θέλουμε όσον αφορά τις συναλλαγές να έχουμε διαφορετικούς ε, κανόνες για τις περιπτώσεις εξαποστάσεως ε, αγοράς. Στη Γαλλία θέλουμε να μην υπάρχει πληρωμή στο υποχρεωτική πληρωμή στο διάστημα δοκιμής του προϊόντος από τον καταναλωτή. Γι' αυτό λοιπόν ο καταναλωτής πρέπει να είναι σε θέση εν πάση ηρεμία να σκεφτεί την αγορά του χωρίς να πρέπει να μπει στις λεπτομέρειες μιας περίπλοκης συναλλαγής ή για το πώς θα αποζημιωθεί στη συνέχεια. Να μην χρειάζεται να πληρώσει. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δύο σημεία επί των οποίων η μέγιστη αρμόνιση όπως προβλέπετε δημιουργεί προβλήματα είναι, εφήγησαν ήδη από την κυρία Καραμαλή. Το πρώτο αφορά τι υποχρεώσει ε, προσυμβατική πριν υπογραφεί το συμβόλαιο τη ενημέρωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει κάτι που μα ικανοποιεί εκτός από το σημείο 9 για την υποχρέωση εκ των προτέρων ενημέρωση, ούτως ώστε ε, να υποχρεούται ο επαγγελματίας να χορηγεί την ενημέρωση και δεν μένει περιθώριο στα κάτι μελη να προσαρμοστούν γιατί προβλέπει μέγιστη εναρμόνιση. Κυρίω ε, να ενημερώνεται σωστά ο καταναλωτή μέσω εμφάνιση των τιμών. Θα πρέπει να εφαρμοστεί εδώ αρχή τη επικουρικότητα. Υπονομεύονται οι εθνικοί κανόνε που είναι αποτελεσματικοί και έχουν παγιωθεί σε εμά όσον αφορά το, το σιδέρωμα, το πρέσεν και του κομμωτέ γιατί να αντικατασταθεί. Ε, η υπονόμευση δεν είναι κάτι σκόπιμο, ε, ε, ούτε είναι υπέρ της εσωτερικής αγοράς, ούτε μιλάμε και για υπερβολικά ποσά. Μετά οι καταχρηστικές ρήτρε. Επί της ουσίας συμφωνούμε με τον ορισμό που προτείνεται, κάτι που ήδη ισχύει, εκτός από την ανεφορά της καλής πίστος, που δεν λέει τίποτα στη Γαλλία και περιπλέκει την κατάσταση. Ε, να παρα μια καταχρηστική ρήτρα δεν δεσμεύει τον καταναλωτή, συμφωνούμε από αυτού. Έχουμε δύο αμφισβητήσεις. Πρώτον, να αποφευγεί κάθε υποχώρηση στον την προστασία στις πρόσωπο με πρόσωπο συμφωνίες, να εντοπίζονται οι καταχρήσεις αν υπάρχουν. Ε, λοιπόν, στις ατομικές ρυθμίσεις θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη και όχι στις προ στα ατομικά συμβόλαια και όχι στα προσυνδεταγμένα συμβόλαια και κάτι που ανέφερε και η συγγήτρια. Ε, ε, οι μαύρες λίστες, οι ρήτρες που, θεωρούνται εν πάση περιπτώσει καταχρηστικές ή να έχουμε λίστες φαιές για αυτές τις ρήτρες που θεωρούνται, υπάρχουν και ασύστονται είναι καταχρηστικές. Ε, αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από τον πολιτισμό που επικρατεί σε κάθε χώρα, την πολιτιστική προσέγγιση. Οι ευρωπαϊκοί κατάλογοι δεν πρέπει να είναι ενιαίοι κατάλογοι που να ισχύουν σε όλες τις χώρες να είναι κοινέ λίστες που θα εφαρμόζονται συμπληρώνοντας τις εθνικές λίστες που είναι συγκεκριμένες και ειδικέ. Και εδώ χαιρετίζω τον νέο συνάδελφο Μία Μπάμπ που εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το βλέπω αυτό με μεγάλη χαρά. Η κυρία Καραμαλή και στη συνέχεια θα ακούσουμε την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ναι, για να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο τμήμα ανταλλαγών, θέλω να έρθω στο θέμα των εγγύσεων. Η μόνη νόμιμη εγγύηση, γιατί εδώ υπάρχουν ε, δύο προβλήματα, το ένα νομίζω βρίσκει σύμφωνες πολλές χώρες, είναι το θέμα του δικαιώματος ε, προσφυγής του καταναλωτή όταν τίθεται πρόβλημα με την εγγύηση. Εδώ πιστεύω ότι το κείμενο είναι άκαμπτο, γιατί μονομερός μόνο ε, μπορεί να ε, ζητήσει είτε την επιστροφή, είτε την αποζημίωση, είτε την επισκευή, ο καταναλωτής πρέπει να έχει την επιλογή. Και το δεύτερο κόλλημα είναι νομικό και έχει να κάνει με την έλλειψη βεβαιότητας ε, για την ισχύ της ε, εγγύησης. Εδώ είναι και θέμα αστικού δικαίου που έχουμε εμείς και που ισχύει σε όλες τις συναλλαγές. Αν εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον έχουμε ευρωπαϊκή οδηγία για μέγιστη εναρμόνιση, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρο σήμερα. Αν παραμείνει η διάταξη αυτή, είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας και είναι κάτι από τα πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Ευχαριστώ. Ήμκο. Μάλκομ. Εδώ ακούσαμε πολλά και διάφορα πράγματα. Δεν μπορούμε βέβαια να απαντήσουμε σε όλα σήμερα το απόγευμα. Σίγουρο οι και οι σκιώδες σα άκουσαν προσεκτικά. Θέλουν κι άλλοι από την Επιτροπή μας εδώ να πάρουν το λόγο και να σχολιάσουν. Τον κύριο έχω πρώτα, κυρία Βερνιό και ο Ρόσφορ. Γάλλοι όλοι. Θα πάρουν το λόγο λοιπόν. Μπορούν να έχουν κι άλλε ευκαιρίε βέβαια να μιλήσουν μαζί σα, αλλά χαίρομαι που θα του ακούσουμε εδώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να χαιρετήσω την πρωτοβουλία του Μάλκομ Χάρμπουρ και του Πιέρ Λεκηγέ. Είναι μια πρεμιέρα στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιτρέπει να ξεκινήσει μια νέα εποχή στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, στην ευρωπαϊκή οικοδήμαση, με καλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων για τη λήψη κοινοτικών αποφάσεων. Όσον αφορά την πρόταση οδηγία, πρέπει να πω ότι διαβάζοντα την έκθεση τη κυρία Καραμαλή, Αισθάνθηκα ήσυχο διότι εντοπίσαμε τι ίδιε δυσκολίε, τι ίδιε αβεβαιότητε και επίση τι ίδιε ενδεχόμενε λύσει. Θα ήθελα απλώ να περιοριστώ σε δύο σχόλια. Εν πρώτη, συμφωνούμε όσον αφορά σκοπιμότητα υπάρξεω του κειμένου. Επίση, συμφωνώ μαζί σα στην Εθνοσυνέλευση και συμφωνεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υπάρχει ένα κείμενο που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών από τη μια πλευρά, βέβαια διατηρώντα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων από την άλλη και πιστεύω ότι χωρί υψηλό επίπεδο προστασία του καταναλωτού δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και χωρί εμπιστοσύνη δεν είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε το διασυνοριακό εμπόριο καθώ και την εσωτερική αγορά. Και πιστεύω ότι εν αυτή τη ενία μπορούμε να συνεργαστούμε για να εντοπίσουμε τα τμήματα τη προτάσεω που κατά την άποψή σα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μέγιστη στοχευμένη εναρμονήσεω όπω είναι οι ορισμοί, ε, το δικαίωμα υπαναχώρηση και απόσυση τη ενδιαφέροντο αγορά. Ε, μπορούμε να επεξεργαστούμε κάποια συγκεκριμένα θέματα που είναι σύμβολο για του Γάλλου καταναλωτέ τη προστασία του καταναλωτού όμω, όπω είναι το θέμα τη νομική εγγύηση και τα κρυμμένα ελαττώματα. Λοιπόν, ε, μπορούμε να βασιστούμε στην άοκνη εργασία του κυρίου Σουβάμπ για να εξευρεθεί κάποια λύση. Και επιτρέψτε μου να σα πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι με τον συνάδελφο Φιλίπ Ζουβέν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να μην δημιουργηθεί το συνέστημα ότι απειλούνται τα διάφορα κεκτημένα δικαιώματα όσον αφορά την προστασία του καταναλωτού σε εθνικό επίπεδο. Και ευχαριστώ και ελπίζω να συνεχίσουμε αυτή τη διαβούλευση. Ευχαριστούμε κύριε Δανιό, έχει το λόγο. Περνάει ο χρόνο, οπότε σύντομα παρακαλώ. Βεβαίω, γιατί και ο συνάδελφο Αμπάντ με κάλυψε σε έναν βαθμό. Λοιπόν, χαιρετίζω και εγώ τους συναδέρφους βουλευτές της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Είμαστε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Επιτέλους, για πρώτη φορά εφαρμόζουμε μια τέτοια διαδικασία. Χαίρομαι λοιπόν που συνεργαζόμαστε και μάλιστα για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Συγχαίρω τη Μαριέτα, η οποία μάλιστα είναι από τη δικιά μου εκλογική περιφέρεια. Διπλά συγχαρητήρια λοιπόν και τον κύριο Λαμπέρ έχω συναντήσει. Πολύ καλά όσα είπε, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Κατά την ε, προεκλογική εκστρατεία σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα στη Γαλλία, ακούσαμε ότι η Ευρώπη δεν προστατεύει αρκετά τους καταναλωτές. 85% όμως της νομοθεσίας έχει να κάνει με την καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Το κείμενο αυτό λοιπόν πρέπει να πετύχει. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλες οι πολιτικές ομάδες για το ότι χρειάζεται το ευρωπαϊκό όραμα. Είναι αναγκαίο και δεν περνάει μέσα από μια μέγιστη εναρμόνιση η οποία θα οδηγήσει σε επαναχώρηση ενδεχομένως στο εθνικό δίκαιο και τις ρυθμίσεις, όχι. Όλοι θέλουμε το ίδιο. Να ισχύσει επικουρικότητα, να προστατευτούν τα δικαιώματα των κρατών χωρών και σίγουρα να μελετήσουμε πολύ καλά ένα θέμα που έχει να κάνει με διάφορε λεπτομέρειε στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Σίγουρα δεν είναι εύκολο με ταξί 27 χωρών, έχουμε όμω τη βούλη σε κατέρωθαν και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ο κύριο Ροσφόρ. Ναι, κοιτάξτε. Τελικά δεν είναι μεγάλο μυστικό που διαπιστώνεται ότι μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Γαλλικού Κοινοβουλίου υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που αφορούν το σχέδιο αυτοοδηγίας δύο απαντήσει να δώσω σε δύο συναδέλφου στο Παρίσι στην κυρία Γκρόμε, που αναφέρθηκε εκτενώς στην πώληση εξ αποστάσεως, να πω ότι είναι ένα θέμα επί το οποίο μπορούμε να εργαστούμε μέσω τροπολογιών για να σεβαστούμε κάποιο πλαίσιο, το μπορεί να βοηθήσει στη μέγιστη εναρμόνιση και εν αυτή περιπτώσει εγώ προσωπικά είμαι υπέρ διαγραφής του τέταρτου εδαφίου σε αυτό αναφέρθηκε, που λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να απόσχουν από την απαγόρευση στα μέρη να εκτελέσουν τι βατικέ του υποχρεώσει κατά τη διάρκεια τη περίοδου υπαναχώρηση, δυνατότητα αλλαγή απόψεω. Μπορούμε να επεξεργαστούμε το κείμενο, βέβαια. Για να απαντήσω στον άλλο συνάδελφο, τα πήγε για τι καταχρηστικέ ρήτρε. Νομίζω ότι καταλαβαίνω αυτά που λέει και αντίθετα πιστεύω ότι από αυτού του θέματο θα είναι δύσκολο να βρούμε κάποια απάντηση όσον αφορά τη μέγιστη εναρμόνιση. Θεωρώ ότι η ελάχιστη εναρμόνιση σίγουρα θα είναι μόνο τρόπο να προχωρήσουμε, διότι ένα κατάλογο είναι χρήσιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σίγουρα είναι χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν λίστα, πρέπει να το ξέρετε. Αντίθετα, θα πρέπει ο καθένα, κάθε κράτο μέλο να μπορεί να έχει προφανώ τη δυνατότητα να έχει αυτέ τι ρήτρε. Στη Γαλλία, επενθυμίζω ότι υπάρχουν 20 καταχρηστικέ ρήτρε στην περίπτωση μίσθωση ακινήτων που είναι στα πλαίσια τη συμβάση και θα πρέπει να γίνουν σεβαστέ. Και δεν πιστεύω ότι η διαδικασία τη επιτροπολογία μπορεί να μα επιτρέψει να επικαιροποιήσουμε πολύ γρήγορα έναν κατάλογο που χρειάζεται να είναι ζωντανό χρονικά. Επ' αυτού ίσω πρέπει να φύγουμε τη μέγιστη εναρμόνιση. Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε μεταξύ μα. Προτείνω κύριε Πρόεδρε να ακούσουμε άλλους δύο ομιλητές από αυτή την πλευρά και μετά να σας δώσω τη σκητάλη για απαντήσεις και μετά θα καταλήξω συμπεράσματα διότι έχουμε μείνει κάπως πίσω. Ο κ. Λέχνερ θέλει να μιλήσει και η κυρία Γκέπχαρτ. Υπάρχει άλλος ο οποίος επιθυμεί να μιλήσει. Από την πλευρά μας ο κ. Λέχνερ πρώτα και μετά η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι στη Γαλλία, δεν είμαι υπέρ της μέγιστης εναρμόνισης ε, όλα εξαρτώνται από το πού θέλουμε εναρμόνιση. Δεν πρέπει να έχουμε απλά μια γενική μέγιστη εναρμόνιση. Αλλά εάν έχουμε πλήρη εναρμόνιση σε κάποιον συγκεκριμένα τομέα, θα πρέπει να φροντίσουμε αυτό να είναι προς όφελος των καταναλωτών. Υπάρχουν, για παράδειγμα, πολλοί Γάλλοι πολίτες ε, από το Στρασβούργο που ψωνίζουν στο ΚΕΛ ή κάποιος ε, Γερμανός μπορεί να ε, αγοράζει πράγματα στη Γαλλία. Και αυτούς τους πολίτες θα τους επωφελούσε μια ευρωπαϊκή λύση για σε κάποιους τομείς, όχι παντού όμως. Καμία Εάν καμία νομική τάξη, ούτε η ισπανική, ούτε η γαλλική, ούτε η γερμανική δεν ε, μπορούν να ε, ε, χωρίσουν κάποια θέματα, τότε δεν θα έχουμε και τίποτα. Γενικά, να προχωρήσουμε με προσοχή. Ευχαριστώ. Και η τελευταία ομιλήτρια, κυρία Κέπχαρτ. Ευχαριστώ. Ήθελα να αναφέρω ένα θέμα που θύχτηκε από τους συναδέλφους στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, το δικαίωμα επαναχώρησης. Δεν, έχουμε, ε, δεν μπορούμε εδώ να έχουμε πλήρη εναρμόνιση, διότι το δικαίωμα επαναχώρησης έχει τόσο διαφορετική μορφή ε, στα διάφορα κράτη-μέλη που θα ε, συναντήσουμε σημαντικές δυσκολίες. Στη Γερμανία ο υπολογισμός της προθεσμίας επαναχώρησης ξεκινάει τη στιγμή που έχει εκδοθεί και το τελικό τιμολόγιο. Ε, στο, σε άλλα κράτη-μέλη ξεκινάει με την παραγγελία. Ε, σε κάποιες χώρες οι προθεσμίες είναι 30 μέρες, σε άλλες είναι 60 μέρες. Είναι τόσο διαφορετικές οι ρυθμίσεις που δεν μπορούμε να τις συνδυάσουμε. Το να πούμε τώρα ότι θέλουμε ενιαίο κανόνα, αυτό σημαίνει ότι στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιταλία θα συναντήσουμε σημαντικές δυσκολίες με τους πολίτες, διότι δεν θα καταλάβουν, θα πούνε ότι... Ε, ότι ε, καταπατώνται δικαιώματα για τα οποία αγωνιστήκαμε. Διότι, να μην ξεχνάμε ότι τα δικαιώματα αυτά υπαναχώρηση είναι δικαιώματα για τα οποία έχουν αγωνιστεί οι πολίτε των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα ενό τομέα όπου δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εναρμόνισης. Δεν λέω ότι δεν θέλουμε καθόλου εναρμόνιση. Εγώ μιλάω για μεικτή εναρμόνιση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σημείο προς σημείο. Πού μπορούμε να το κάνουμε αυτό και πού όχι κυρία Τούρνεν μου ζήτησε να, τη δυνατότητα για μια τελική παρατήρηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους Γάλλους συναδέρφους. Ε, βρίσκω ότι ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση σήμερα. Ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε παραδείγματα γαλλικά προβλημάτων, διότι είναι σημαντικό όταν εμεί εδώ εκπονούμε νομοθεσία που θέλουμε να καλύψει όλα τα θέματα, να ακούσουμε τα εθνικά ε, προβλήματα και όχι μόνο τη Γαλλία, όλων των κρατών μελών. Ε, θα σας παρακαλούσα να μας στείλετε τα προβλήματα αυτά ε, για να συμβάλλετε στη νομοθετική μας διαδικασία. Και επίσης ε, θα ήθελα συλλογισμούς από εσά για τη σχέση ανάμεσα στη νομοθεσία που εκπονούμε εδώ πέρα και το δικό σας ενοχικό δίκαιο αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Νομίζω ότι θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια της διαδικασίας. Ελπίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε ανταλλαγές απόψεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέρφους. Ε, κύριε Πρόεδρε, σας δίνω το λόγο για να ακούσουμε τις ε, τελικές παρεμβάσεις της ομάδας σας. Ε, θα δώσω το λόγο στον Κριστόφ Καράς και μετά ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τους δύο εισηγητές μας. Σφαπ και Καραμαλή. Οπότε, ο Κρίστο Καές πρώτα από τους σοσιαλιστές. Ναι, δύο παρατηρήσει για τη συζήτηση που έγινε. Πρώτα απ' όλα δεν έχω την αίσθηση ότι τα προβλήματα που βάζει η Γαλλία είναι προβλήματα που διακρίνουν μόνο τη Γαλλία. Και άλλε χώρε έχουν τα ίδια προβλήματα και άλλε οργανώσει τα θέτουν. Είναι ευρωπαϊκά προβλήματα, δεν είναι εθνικά προβλήματα δηλαδή. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, και εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ θετική η συζήτηση, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί παρετέρω το θέμα της μέγιστης εναρμόνισης. Εμείς δεν τη θέλουμε. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο έχουμε καταλήξει. Γιατί πλήττει τα δικαιώματα των καταναλωτών ακριβώς. Καλύτερα μια ελάχιστη εναρμόνιση υψηλού επίπεδου παρά μια ανώτατη μέγιστη εναρμόνιση που είναι όμως χαμηλού επίπεδου μίλησε ο κύριο Σβάμπ για στοχοθετημένη εναρμόνιση. Εντάξει, αυτή είναι μια νέα έννοια, ενδιαφέρον στοιχείο. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, εμείς δεν θέλουμε μία εναρμόνιση η οποία να πλήττει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ευχαριστούμε. Τώρα, Μαριέτα Καραμαλή και μετά ο κύριο Βάμπ. Ναι κύριε Πρόεδρε, για να κλείσω κατά κάποιο τρόπο το πρώτο στάδιο, θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να επενθυμίσω ότι εν τέλει όσον αφορά την ανάγκη εναρμονίσεως του δικαίου του, όσον αφορά την κατανάλωση στην εσωτερική αγορά να κάνω ένα σχόλιο. Στη Βόρεια Αμερική υπάρχει πλουραλισμός νομοθεσίας. Αυτό δεν εμπόδισε την ύπαρξη εσωτερικής αγοράς. Και διαπίστωσα ότι μέσω των διαφόρων τοποθετήσεων των Ευρωβουλευτών η άποψη των Γάλλων είναι κάτι που το μοιράζονται και άλλες χώρες και διάφορες διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Να επενθυμίσω όσον αφορά το, την ομοθεσία για την κατανάλωση όπως προτείνεται υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, καλύτερη εγγύηση όσον αφορά την εξοπιστία των προϊόντων χρειάζεται πιο βιώσιμα προϊόντα να παράγονται. Και στο ψηφιακό τομέα τα διάφορα προϊόντα που πολλούνται και πολιτιστικά προϊόντα που πολλούνται πρέπει να καλύπτονται. Λοιπόν, λέγεται ότι οι νόμοι θα πρέπει να, κάνουν, να υποφέρουν οι ανισότητες. Εδώ έχουμε τις ανισότητες μεταξύ των διαφόρων καταναλωτών των χωρών αλλά και των διαφόρων ατόμων που δεν γνωρίζουν τον νόμο, τα δικαιώματά τους. Και παίζουν οι επαγγελματίε με τα δικαιώματά τους. Πριν προχωρήσει ο προβληματισμός, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να κάνουμε με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη δράση των διαφόρων ομάδων. Χρειάζεται να επεξεργαστούμε τους ορισμούς και τους όρους υπαναχωρήσεως ε, και υπ' αυτού του όρου να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση. Ο κύριο Σβάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Εισηγήτρια. Έχω ήδη πει ότι η εσωτερική αγορά και η προστασία των καταναλωτών είναι δύο πλευρές ε, του ιδίου νομίσματος. Ε, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μα ότι η εσωτερική αγορά θα έχει περισσότερο δυσνοριακό εμπόριο εάν καταφέρουμε να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα μαζί σας στο θέμα αυτό. θα πρέπει να προωθήσουμε ακριβώς τη βάση της Ευρώπης. Θα πρέπει δηλαδή να προωθήσουμε το εσωτερικό εμπόριο όχι μόνο για ε, τις... Ε, ε, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Είδαμε τι συνέβη στην οδηγία για τις καταναλωτικές πιστώσεις. Ε, τα κράτη-μέλη είπαν ότι είμαστε υπέρ της ε, πλήρους εναρμόνισης στο σημείο 1 και στο σημείο 2 βλέπουμε 27 εξαιρέσεις διότι στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία κλπ. Ε, υπάρχει και το εθνικό δίκαιο. Αυτό δεν έχει νόημα για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες και του καταναλωτέ. Χρειάζονται διαφάνεια, σαφήνεια, απλά νομοθετικά κείμενα και γι' αυτό η εναρμόνιση σε κάποιους στοχευμένους τομείς έχει νόημα μόνο όταν είναι σαφής. Και πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να επηρεάσουμε το Συμβούλιο ώστε να καταλήξει σε απλές κατανοητές λύσεις. Η τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι υπάρχει μια μακρά σειρά γαλλικών ε, φορέων που αναφέρθηκαν που υπάρχουν όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και σε πολλά άλλα κράτη-μέλη και ε, πιστεύω ότι είναι θέματα που θα πρέπει να εξετάσουμε. Για παράδειγμα, στις δημοκρασίες στο διαδίκτυο στα διαδίκτυα, ε, σε ηλικιακά καταστήματα. Θέλουμε στους τομείς αυτούς να βελτιώσουμε την προστασία των καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν θα βλάψει κανέναν. Το άλλο θέμα είναι ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν ε, κάποιες εξελίξεις ε, στην Ευρώπη που όχι θα, θα δυσκολέψουν το διασυνοριακό εμπόριο. Έχουμε τον κανονισμό Ρώμη 2 ε, ε, ε, της Βασιλείας κλπ. Έχουμε την περίπτωση Άλπενχοφ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά και επικοδομητικά να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για τους Ευρωπαίους πολίτες. Λύσεις που να μπορούν να καταλάβουν οι πολίτες. Ίσως θα ήταν χρήσιμο στο μέλλον να έχουμε άλλη μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάντω για τις πολύτιμες παρατηρήσεις σας. Πρόεδρε, εσείς για το τελικό συμπέρασμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Μάλκομ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ θερμά όλους. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να οργανωθεί αυτή η κοινή συνάντηση που πραγματικά συμβαίνει για πρώτη φορά. Το έργο αυτό, όπως είπε και ο κύριος Βά πολύ σωστά, πρέπει να συνεχιστεί. Και φυσικά και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας. Όπως όμως διαπιστώσατε, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των εθνικών ε, βουλευτών, τόσο ε, του κυβερνητικού σήματος όσο και της αντιπολίτευσης, και όπως είπε ο κύριος Σφαπ και ο Κριστόφ Καράς πριν από λίγο, δεν πρόκειται για γαλλική θέση όμως, πρόκειται για θέση που πιστεύω έχουν και άλλες χώρες. Δηλαδή να μην κάνουμε πίσω, το είπαν αυτό πολύ όσον αφορά τα σημερινά δικαιώματα των καταναλωτών. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και τέλος, η, η εναρμόνιση, η μέγιστη εναρμόνιση στοχοθετημένη, επαναλαμβάνω αυτή την έκφραση, στοχοθετημένη να εφαρμόζεται με ρεαλιστικό τρόπο. Αυτό είναι αναγκαίο. Το μελλοντικό κείμενο λοιπόν θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ευρωπαίων καταναλωτών. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά ε, για αυτήν την συνάντηση που γίνεται για πρώτη φορά και ελπίζω να επαναληφθούν και άλλες τέτοιες συναντήσεις. Μάλκομ. Να σε ευχαριστήσω, Πιέρ, και να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέρφους σου για τη συνεισφορά τους. Ως Βρετανός ε, πολιτικός ε, ενδιαφέρομαι και εγώ, όπως και εσύ, ε, για πρακτικές λύσεις και από αυτήν την άποψη νομίζω ότι εργαζόμαστε σκληρά στην Επιτροπή μας ε, για να καταλήξουμε σε έναν λογικό συμβιβασμό. Ε, νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Ε, πραγματοποιήθηκε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν και από τις δύο πλευρές και στο Παρίσι και εδώ στις Βρυξέλλες που ε, καταφέρανε να ανταμάσουν ε, την τεχνολογία. Ο πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά τους διερμηνείς Πιστεύω όμως, συνεχίζει ο Πρόεδρος, ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερες ε, σύντομες και επικεντρωμένες ανταλλαγές απόψεων. Μία ώρα εργαστήκαμε μαζί. Ε, ήταν ε, ιδιαίτερα παραγωγική η εκδήλωση αυτή. Ελπίζω να έχουμε και στο μέλλον άλλες ευκαιρίες να το κάνουμε αυτό. Σήμερα είχαμε εδώ συνάντηση με βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια, 21 βουλευτές παραβρέθηκαν για να συζητήσουμε την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Ε, ήταν λοιπόν ένα καινοτόμο απόγευμα από τη δική μας πλευρά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας ε, και κλείνω την ε, σύνδεση με το Παρίσι. Κλείνω και την ε, διάσκεψη ευχαριστώντας και εσάς και τους συναδέλφους μου. Πολύ καλό βράδυ από τις Βρυξέλλες. Μάλκομ. Μάλκομ. Μάλκομ. Μ' Μάλκομ. Ήθελα να πω ότι ναι, είμαι ρεαλιστής και υπέρ των πρακτικών λύσεων, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι είμαι από Αγγλίδα μητέρα, ε, που γεννήθηκε στην Ολλανδία, οπότε καταλαβαίνεις.